Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε γιατί είναι γεμάτη η ημερήσια διάταξη. Ξεκινάμε με το πρώτο θέμα. Θέλω να σας ενημερώσω πως υπήρχαν αιτήματα να αλλάξει η ημερήσια διάταξη της σημερινής και αυριανής συνεδρίασης. Το πρώτο θέμα το έθεσε ο κύριος Μποστινάρου, ο οποίος λόγω άλλων υποχρεώσεων θα λείπει μεταξύ 3 ε, και 4 και 4. Γι' αυτό ζήτησε να ψηφίσουμε κάποια στιγμή κατά την οποία θα είναι παρόν. Νομίζω πως έχουμε τόσα πολλά πράγματα να ψηφίσουμε ώστε μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι και άρα προτείνω να δεχτούμε το αίτημα του Βίκτορα. Ένα δεύτερο θέμα είναι επίσης μια τυπική αλλαγή γιατί βλέπετε πως έχει έρθει ο κύριος υπουργό Ανδρέας Παυρογιάννης οπότε προφανώς ε, τώρα θα γίνει η ανταλλαγή απόψε με τον κύριο Υπουργό ναι, την ε, Κυπριακή Προεδρία και τον ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, τον κύριο Μαυρογιάννη. Αμέσως δηλαδή με τα, τα τυπικά θα μιλήσουμε με τον κύριο Υπουργό, κάτι το οποίο σημαίνει πως τα σημεία 4, 5 και 6 της ημερήσιας διάταξης θα τα δούμε την Πέμπτη από τις 9 μέχρι τις 10.30. Ορίστε. Αυτό προτείνω λοιπόν για την ημερήσια διάταξη. Ο Μάρκος Πίπερ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε για την ψηφοφορία θα ήθελα να μιλήσω τη σημερινή σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε τις πέντε εκθέσεις που ασχολούνται με τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2014-2020. Με συγχωρείτε, λέει πρώτος, ακούτε εσείς αγγλικά. Υπάρχει μια τελείως διαφορετική γλώσσα στο κανάλι 2, λέει πρόεδρος, αλλά όχι τα αγγλικά. Υπάρχει διερμηνία τώρα στα αγγλικά, ωραία. Λοιπόν, Μιλάμε λοιπόν για τις βασικές κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Διαρθρωτικής Πολιτικής 360 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους τις τελευταίες μέρες και νύχτες δούλευαν όλο το 24ωρο για να υποβάλουν ε, καταλόγους ε, ψηφοφορίας. Γνωρίζω και ο ίδιος αυτές τις ε, διαδικασίες, αλλά ως απλό μέλος πρέπει να πω το εξής. Χτες, 3 η ώρα το απόγευμα, είχα για πρώτη φορά την δυνατότητα να δω τις ε, συμβαστικές προτάσεις και να τις συζητήσω με το κόμμα μου. Χτες, 3 η ώρα το απόγευμα και μάλιστα ε, μου είπαν οι συγητές πως αυτές είναι οι συμβαστικές προτάσεις, δεν μπορείτε να αλλάξετε τίποτα και πρέπει να τις δεχτείτε. Ε, και αναρωτιέμαι, ποια πιθανότητα ε, έχω εγώ ως μέλος της Επιτροπής μας να παρέμβω επιπλέον. Δεν υπήρχε καν ο κατάλογος της ψηφοφορίας. Μέσα στη νύχτα δε, τρεις ώρα το πρωί, τρεις η ώρα το πρωί μας έστειλε το κατάλογο της ε, ψηφοφορίας. Κυρίε και κύριοι, αυτή η διαδικασία που μας επιβλήθηκε από ολίγους είναι αντιδημοκρατική, δεν είναι διαφανής, είναι αντίθετα σε κάθε κανόνα του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω ε, να ψηφίσουμε σήμερα μόνο τις εκθέσεις εκείνες τις οποίες μπορέσαμε να συζητήσουμε αναλυτικά. Να σου πω επί της ουσίας, δεν συμφωνώ πολλά πράγματα που υπάρχουν σε αυτές τις εκθέσεις, αλλά τουλάχιστον είχαμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Θέλω λοιπόν συγκεκριμένα να ζητήσω το εξή, να ψηφίσουμε σήμερα μόνο το Ταμείο Συνοχής, τι μεθοριακές περιοχέ, δεν θυμάμαι ακριβώ τον τίτλο, ξέρετε τι εννοώ, εκεί που είναι σκιώδηση η Μαρή Τερέζ ε, Σάντσε και την ε, έκθεση του Γιώργη Τσέλερ. Να αναβάλουμε όμως την έκθεση Γιάν Ουλμπριχτ και να αναβάλουμε τον Γενικό κανονισμό για τα διαρθρωτικά ταμεία, δηλαδή την έκθεση Φανίστελ Ρόι. Και λοιπόν, κυρίε και κύριοι, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, τόσο ή άλλως δεν συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα. Και οπωσδήποτε κάτι θα κάνει και η Κυπριακή Προεδρία. Αλλά θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα με την ησυχία μας, να τα διαβάσουμε και να έρθουμε από τις διακοπές και να διαπραγματευτούμε σοβαρά και να έχει και ο απλός βουλευτής τη δυνατότητα να λάβει μέρος. Σας παρακαλώ να δεχτείτε αυτή την αναβολή και θα ήθελα την στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, Marcus, very much. Ε, Ευχαριστούμε, Μάρκους Κωνσταντσε ε, Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να διαφωνήσω με τον Μάρκους Πίπερ και να προβάλλω μια αντίρρηση. Από πέρσι, από τα μέσα Οκτωβρίου, πάρα πολύ εντατικά συζητούμε εδώ το θέμα και για το γενικό κανονισμό. Ως εισηγητέ είχαμε διάφορα έγγραφα εργασίας υποβάλει, τα οποία επίσης συζητήθηκαν εντατικά, όχι μόνο στην ε, Επιτροπή αλλά και στην ομάδα εργασίας και φυσικά και προφανέστατα ε, στις ομάδες ε, εργασία των πολιτικών ομάδων. Στην Επιτροπή εδώ έχουμε συζητήσει επανειλημμένα ενδεχόμενες συμβαστικές προτάσεις και οι συμβαστικές τροπολογίες που υποβάλλουμε οι συγητές είναι αποτέλεσμα αυτής της μακράς συζήτησης διαφανής και εκτενής ε, και εδώ και στις ομάδες εργασίας. Πιστεύω ότι θα ε, διαπράταμε τεράστιο σφάλμα εάν σήμερα δεν ε, σφραγίζαμε με ψηφοφορία ε, την επιτυχία ε, αυτή τη προσπάθεια που μα δίνει και την εντολή για διαπραγματεύσει. Θα ήμασταν η πρώτη επιτροπή που σε ένα μεγάλο πακέτο πολλών διαφορετικών προγραμμάτων, έργων σχεδίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψήφιζε και θα είχαμε και διαπραγματευτική εντολή. Γι' ε, αυτό είναι σημαντικό μήνυμα και μάλιστα πολιτικά σημαντικό μήνυμα του Κοινοβουλίου προς τα έξω για να διατρανώσουμε ότι με την πολιτική συνοχή έχουμε ένα μέσο στα χέρια μας και ένα εργαλείο για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη να εξέλθουν από αυτή τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και κρίση. Δίνουμε μήνυμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νοιάζεται και ασχολείται με τους πολίτες της περιφέρειες. και είναι σημαντικό να ψηφίσουμε σήμερα. Δίδεται εντολή στους διαπραγματευτές για τον τριμερή διάλογο και πάντα θα ερχόμαστε να το συζητούμε στην Επιτροπή μας εδώ μαζί σας, ενδεχομένως και με μια αλλαγή της διαπραγματευτικής εντολής και η διαδικασία θα εξακολουθήσει να είναι και διαφανής και συναδελφική και σας παρακαλώ να μην επιτρέψετε αυτό το αίτημα ε, του κυρίου Πίπερ να ευδοκιμήσει. Ευχαριστώ, η Πρόεδρος. Ο Φρανσουά Αλφονζή. Oui, euh, nous partageons les, les remarques. Εγώ συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου, της κυρίας Κρέλ. Η εργασία ήταν πολύ εντατική αλλά και δημοκρατική. Μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον συγκητή μάλιστα που έδειξε μεγάλη διαθεσιμότητα και δούλεψε πολύ σκληρά. Πιστεύω πως η Επιτροπή μας έχει κάθε συμφέρον να ψηφίσει γρήγορα και να είναι μάλιστα η πρώτη που θα θέσει σε αυτές τις προτάσεις, διότι καταρχήν αυτός είναι ο ρόλος μας και η ε, και, η αποστολή μας και έπειτα θα πρέπει να δώσουμε, ε, να ενισχύσουμε το τριμερή διάλογο και να έχει το χώρο που χρειάζεται εφόσον η συνθήκη της Λισαβόνας τον έχει ενισχύσει. Εμείς θέλουμε λοιπόν να ψηφίσουμε. Uh, thank you very much. Any other comment on this? Uh, I, don't know if there is a need to... Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ε, να ψηφίσουμε τώρα, γιατί ε, νομίζω ότι είναι η αίσθηση της πλειοψηφίας να παραμείνει στην ημερησία διάταξη και να ψηφίσουμε. Ή θέλετε να, θέλετε να ψηφιστεί το έτοιμά σας τυπικά. Ναι, ο κύριος Πίπερ θέλει να υποβληθεί σε ψηφοφορία το έτοιμά του. Ε, να το πω θετικά τότε. Ποιος θέλει να παραμείνει η μερίσια διάταξη ως έχει, δηλαδή να διεξαχθεί η ψηφοφορία ε, για τις τροποποίησεις των κανονισμών. Ιδού, νομίζω ότι είναι Πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Κατά τώρα. Three votes. Τέσσερις ψήφοι κατά. Οπότε είναι σαφής η πλειοψηφία και η απάντηση. Εγκρίνουμε λοιπόν το στην ε, ημερησία διάταξη και σας θυμίζω ότι ε, ως συνήθως ε, η συνεδρίαση του μεταδίδεται απευθεία στο διαδίκτυο. Για παίρνουμε στο επόμενο θέμα, έγκριση των πρακτικών τη συνεδριασης 29 η και 30 η Μαου. Ω συνήθω σας έχουν διανεμηθεί τα πρακτικά και θα θεωρούν εγκεκριμένα στο τέλο τη συνεδρίασης αν δεν προβάλλει κανεί καμία αντίρρηση. Σημείο 3, ανακοινώσει τη Προέδρου δεν έχω να σα κάνω. Οπότε και μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο επόμενο θέμα στη μερίσια διάταξη που είναι το σημείο 17 ανταλλαγή απόψεων με την Κυπριακή Προεδρία. Ε, τώρα έφτασαν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, έχουμε μα τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ. Η Προεδρία σας θα είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για για την Περιφερειακή Επιτροπή εδώ, αλλά και για πάρα πάρα πολλούς ενεχομένους και δικαιούχου της πολιτική αυτής που περιμένουν να οριστικοποιηθούν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει και για τον προπολογισμό αλλά και για το κανονιστικό πλαίσιο. Σα παρακαλώ να μην λησμονείτε τη ε, σημασία που έχει αυτό ε, και θα πρέπει να το αποδείξει και η Κυπριακή Προεδρία. Έχετε μέσα στο λόγο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Χούμπνερ, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, κύριε και κύριοι. Καταρχήν, επιτρέψατε μου να εκφράσω την ε, ευγνωμοσύνη μου για την πρόσκλησή σας σε αυτή τη συνεδρία. Είμαι ευτυχής ε, που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, ιδιαίτερα σε σχέση με την συνοχή. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλες τις επιτροπές του για το σημαντικό ρόλο που παίζει στην προστασία και πρόθεση του εκδημοκρατισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ενεργού συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων και χάρη στις θεσμικές βελτιώσεις που έγιναν μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Θα ήθελα να σας πω ότι για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας βασικός εταίρος, ότι η Προεδρία μας βασίζεται σε εσά για να προωθήσει το δικό μας όραμα και για να επιτύχει τους κοινούς μας στόχους. Πιστεύουμε σταθερά πως μια ομαλή και επικοδομητική συνεργασία με, την Ευρωπαϊκή, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επιτακτική ανάγκη για να προχωρήσει η Ένωση. Αρκετές ε, συνεδριάσεις έχουν ήδη γίνει, συναντήσεις ανάμεσα στις επιτροπές του Κοινοβουλίου και τους αρμόδιους υπουργούς της Κύπρου, ενώ η διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών το περασμένο Μάιο μας, μας χρησιμεύσε ως οδικός χάρτης για τη συνεργασία μας, αλλά ε, καθώς επίσης ε, η επίσκεψη της διάσκεψης των Προέδρων στην Κύπρο. Από πλευρά μα είμαστε δεσμευμένοι για να προχωρήσουμε σε ενίσχυση αυτή τη συνεργασία και συντονισμό με το Ευρωκοινοβούλιο μέσω μιας διαρκούς ανταλλαγής απόψεων ε, περί των εξελίξεων έτσι ώστε να έχουμε πραγματική πρόοδο για την ατζέντα που έχουμε ενώπιόν μα Γνωρίζετε ότι διανύουμε μία από τις πιο σημαντικές περιόδου της εθνικής μας ιστορίας και για μας τον αναλάβουμε πριν από μία εβδομάδα την Προεδρία του ε, Συμβουλίου είναι υψής της σημασίας. Για πρώτη φορά από την προσχώρησή μας είναι μια μεγάλη πρόκληση αλλά και μοναδική ευκαιρία για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Φυσικά η συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας σε μια κρίσιμη στιγμή καθιστά αυτή την πρόκληση ακόμα πιο απαιτητική. Και επίσης λαμβάνοντας υπόψη πως έχουμε επιτάπητο στι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το δημοσιονομικό πλαίσιο που θα καλύψει την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλίων για την επόμενη προγραμματική περίοδο όπου όλα αυτά συμβαίνουν ε, στη διάρκεια μιας βαθιάς κρίσης με μεγάλες επιπτώσεις στις οικονομίες και την κοινωνία της Ευρώπης ε, καθώς επίσης ε, το γεγονός ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει σοβαρά επηρεάσει τους Ευρωπαίους πολίτες, ενώ η Ευρωζώνη φέρει την τεράστια πίεση. Πρέπει ωστόσο να συνεργαστούμε ώστε η Ευρώπη να αναδυθεί ισχυρότερη από αυτή την κρίση και να εδραιώσει και πάλι τη θέση της στο διεθνές προσκήνιο. Πιστεύουμε πως ε, ε, έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι σημερινές προκλήσεις και να υπάρξει ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή θα είναι το να στηρίξουμε τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσης. Επί τη βάση αυτών των αρχών, ο βασικός στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι να προωθήσει την ιδέα της, εργα... της ε, εργασίας προς μια καλύτερη Ευρώπη μέσα στο πλαίσιο της πρόθεσης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που να είναι πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο. Μια πιο ουσιαστική ένωση που θα συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης με ισχυρότερη δέσμευση για την πρόθεση της συνοχής και της, ε, της και ιδιαίτερη ε, έμφαση στην ε, καταπολέμηση της ανεργίας των νέων έτσι ώστε να κληροδοτήσουμε μια καλύτερη Ευρώπη στις επόμενες γενναίες. Γενικό, το γενικό μας στρατηγικό πλαίσιο και ο στόχος ε, εργασίας προς μια καλύτερη Ευρώπη προωθείται μέσω τεσσάρων βασικών προτεραιοτήτων της Κυπρικής Προεδρίας. Η πρώτη είναι η πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη. Δεύτερον, η Ευρώπη με καλύτερη απόδοση και ανάπτυξη ανάπτυξη στην οικονομία. Τρίτον, πιο κοντά στους πολίτες της με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή. Και τέταρτη προτεραιότητα είναι η Ευρώπη στον κόσμο, πιο κοντά στους γειτονές της. Θα ήθελα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην πρώτη προτεραιότητα της Κυπριακή Προεδρίας, δηλαδή την προώθηση μια πιο αποτελεσματικής και βιώσιμης Ευρώπης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βασικό στόχος της Ευρωπαϊκής Προεδρίας θα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, περί του επόμενου πολιετές δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 η επιτυχής διαχείριση αυτού του ε, θέματος του ΠΔΠ είναι το πιο σημαντικό έργο που έχουμε μπροστά μας και είναι και το σημαντικότερο θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Κυπριακή Προεδρία τους επόμενους 6 μήνες. Το ΠΔΠ είναι ένα βασικό ε, εργαλείο για την οικοδόμηση του μέλλοντος. Ε, σύμφωνα με τα απορίσματα του Ιουνίου, του Συμβουλίου μάλλον του Ιουνίου, θα επιμείνουμε στα αποτελέσματα που επέτυχε η Δανική Προεδρία. Θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Πρόεδρο της Επιτροπής και φυσικά θα συνεργαστούμε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σεβόμενοι το ρόλο του όπως αυτός ορίζεται από τη συνθήκη. Θέλουμε λοιπόν να ε, συμβάλλουμε και να εργαστούμε προς την επίτευξη του στόχου μιας καλύτερης Ευρώπης. Η πρόταση της Κομισιόν έχει δώσει ένα μια πολύ καλή βάση για την έναρξη των προματεύσεων που γίνονται, όπως έλεγα και, παλιό, και προηγουμένως, μέσα σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ε, προβλέψει τους κατάλληλους πόρους ώστε να μπορέσουμε να εξέλθουμε της οικονομικής κρίσης και ε, προμηθεύοντας μια, βάση, μια βάση, σταθερή βάση για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ε, ε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε έτσι ώστε οι δαπάνες να αφιερωθούν σε προγράμματα πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας εφόσον όταν προγραμματίζονται όλα αυτά, όλες οι βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν το δυναμικό για να βοηθήσουν, να προωθήσουν την ανάπτυξη. Ε, παιδεία, καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη θα συμβάλλουν στην στο μακρόπνο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δώσουν και κίνητρα για την ανάκαμψη θα πρέπει να διατηρηθεί μέσα σε όλα αυτά και η αρχή της αριστείας. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολυνθούν, να συμμετέχουν και να μπορέσουν να, ε, να ε, υλοποιήσουν τις, ε, τους στόχους της Ευρώπης 2020. Αποτελεσματική και αποδοτική Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν εν γέννη θα είναι ο στόχος, με στόχο να δώσει όθηση στην, στην απασχόληση ιδιαίτερα για τους νέους. Ο ευρωπαϊκός Προπολογισμό θα πρέπει να έχει τα απαραίτητα μέσα ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους του 2020 ε, με σεβασμό στην αρχή της αλληλεγγύης ε, και με συμβολή στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Ταυτόχρονα οι μηχανισμοί εφαρμογή θα πρέπει να απλοποιηθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί σε σχέση, πάντοτε σε σεβασμό ε, της αρχής της αναλογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό η η πολιτική συνοχή δεν είναι μόνο μια ένδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, αλλά μια ε, σπουδαία επενδυτική πολιτική με σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι επίσης σημαντική πολιτική για την Ένωση που ε, μεριμνεί για τα ευρωπαϊκά αγαθά και εφαρμόζει διάφορες περιβαλλοντικές διατάξεις. Η ε, διατύπωση αυτών των πολιτικών με εστίαση στα αποτελέσματα και στις ποιοτικέ επενδύσεις ε, θα μας ε, βοηθήσει να, να παίξουμε σημαντικό ρόλο και να προωθήσουμε την ανάπτυξη. Η εξέβρεση της σωστής ισορροπίας ανάμεσα στην πλευρά των ε, δαπανών και των εσόδων είναι πολύ σημαντική και μέσα στη πτυχή των δαπανών θα πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα στοιχεία και τις διάφορες πολιτικές. Φυσικά, εξίσου σημαντικές είναι οι βασικές αρχές της, της δικαιοσύνης και της ισότητας ανάμεσα στα κρατη και πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας όταν ε, μιλάμε για τις ε, συμβολές των, τις φορές, συνεισφορές συγγνώμη, των κρατών μελών στον προϋπολογισμό. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα εργασία μας, το ΠΔΠ θα είναι στην ημερήσια διάταξη όλων των συμβολίων γενικών υποθέσεων υπό την Κυπριακή Προεδρία μέχρι ότου να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει Επιπλέον ε, των ε, επισήμων ε, συνεδριάσεων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων θα γίνει και μια άτυπη συνεδρίαση στα τέλη του Αυγούστου στην Κύπρο για το, από, το Υπουργείο, από τους Υπουργούς ε, Εξωτερικών για να συζητηθεί ε, το ΠΔΠ. Ξεκινώντας από χτες, ξεκινήσαμε εντατικέ διμερείς ε, επαφές με όλα τα κρατημέλη, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτών των επαφών. Θα προχωρήσουμε επί τη βάση του διαπραγματευτικού κούτιου το οποίο θα το αναπτύξουμε περαιτέρω, σύμφωνα και με τις εξελίξεις των συζητήσεων στο Συμβουλίο. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία συνδέεται ε, στενά και η διαπραγματευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε μια συνάντηση, μια σύσκεψη πριν από κάθε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και μια ενημέρωση μετά από κάθε Συμβούλιο. Πρόθεσή μας είναι να ολοκληρώσουμε το διαπραγματευτικό κουτί πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας μας, ένα αναθεωρημένο διαπραγματευτικό κουτί θα συζητηθεί το Σεπτέμβριο σε επίπεδο Κορεπέρ και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 24 Σεπτεμβρίου. Φυσικά στόχος μας είναι να μπορέσουμε να, να προχωρήσουμε σε ορίμανση του θέματος ώστε να φτάσουμε σε μια πρώτη πολιτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το Οκτωβρίου. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στο επίπεδο κορεπέρα ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για το Δεκέμβριο. Οι διαπραγματεύσεις βέβαια γίνονται παράλληλα με εκείνες που γίνονται για τα, τις διάφορες τομεακές πολιτικές που καλύπτονται από το πί Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο, ενώ ταυτόχρονα δεν θα προκαθορίσουμε το αποτέλεσμα των συζητήσεων για το πι δελτα πι. Θα έχουμε μια μερόληπτη προσέγγιση και όσον αφορά την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε την ίδια διαδικασία ώστε να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγματευτική ε, διαδικασία. Όπως σας έλεγα, αυτή ήταν η πρακτική που ακολουθήθηκε και με την προηγούμενε τις προηγούμενες την Πολωνική και την Δανέζικη. Η Προεδρία επίσης θα ενημερώσει το, θα ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για την έκβαση των συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο στόχος μας είναι να ενισχυθεί, να εντατικοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο, ενώ θα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ώστε να ε, διευκολύνουμε και να εξασφαλίσουμε την συγκατάθεση του Κοινοβουλίου στο πακέτο, για το πακέτο εγκαίρως και έτσι ώστε να επιτύχουμε την υιοθέτηση, την έγκαιρη υιοθέτηση ε, των απαραίτητων αποφάσεων. Θέλουμε να δουλέψουμε σκληρά και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο. Το αναγνωρίζω ότι είναι φιλόδοξο. Υπάρχουν πολλέ παράμετροι που εμπλέκονται σε αυτέ τι διαπραγματεύσει, ορισμένε πέραν του ελέγχου μα. Αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει σωστά αυτή η δουλειά ε, προ όφελο των κρατών μελών και της Ένωσης ε, εν γέννη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, επιτρέψατε μου να πω δύο λόγια για τις προτεραιότητές μας σε σχέση με τη νέα πολιτική συνοχής. ενώ διατηρείται ο στόχο για την οικονομική και κοινωνική συνοχή επί τη βάση τη θεμελιώδου αρχή της, συνοχής, αλληλεγγύης, η συνοχή αποτελεί ένα κλειδί για την προώθηση των επενδύσεων, την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόληση, καθώς και τη διενέργεια διαρθρωτικών αλλαγών σε ολόκληρη την Ένωση. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων μας, όπως αυτοί προβλέπονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και όσον αφορά την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς. Ε, θέλουμε να έχουμε μια πιο αποτελεσματική πολιτική λοιπόν και αυτό το όραμα αντικατοπτρίζει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο για την περίοδο 2014-2020. Σε αυτό το πλαίσιο, μια από τις βασικές προτεραιότητες της ε, Κυπριακής Προεδρίας είναι να διευκολύνει την έγκαιρη συμφωνία για το νέο νομοθετικό πακέτο για την πολιτική συνοχή. Τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες χρειάζεται να προετοιμαστούν αρκετά νωρί για τη νέα προγραμματική περίοδο ώστε να ξεκινήσουν ομαλά την εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. Γι' αυτό το λόγο, ως Προεδρία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ε, ώστε να επιτύχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, στο Συμβούλιο έχει γίνει μεγάλη πρόοδος κατά τη διάρκεια της Δανέζικης Προεδρίας. Ένα σημαντικό τμήμα της νομοθεσίας αυτής ε, έχει προσωρινά συμφωνηθεί σύμφωνα με τους κοινού μας στόχους για απλοποιημένη και αποτελεσματική πολιτική. Ωστόσο, μένει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει. Η Κυπριακή Προεδρία έχει ήδη ξεκινήσει εντατική δουλειά στο Συμβούλιο με στόχο να ολοκληρώσει να όλα τα εκκρεμή ζητήματα μέχρι το τέλος του 2012. Η πολιτική συνοχή θα συμπεριληφθεί στην ατζέντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων του Οκτωβρίου και του Δεκεμβρίου χρειάζεται να φτάσουμε σε συμφωνία επί τη βάση της γενικής προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση των έλεγχων, την δημοσιονομική διαχείριση, το κοινό στατικικό πλαίσιο, την εδαφική ανάπτυξη και άλλα εκκρεμή ζητήματα. Ταυτόχρονα αποδίδουμε με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο. Καλωσορίζουμε και εκτιμούμε τις σπουδαίες προσπάθειες που έχουν γίνει από την Επιτροπή σας που έχουν οδηγήσει στις σημερινέ και στις αυριανές από ό,τι κατάλαβα ψηφοφορίες για τις ε, ε, αντίστοιχε εκθέσεις σχετικά με το νομοθετικό πακέτο περί για ε, την περίοδο 2014 με 2020. Βασιζόμενοι στα αυτά που έχουν ήδη επιτευχθεί στο Συμβούλιο, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε μαζί σας και να μπορέσουμε έτσι να προχωρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο για το θέμα αυτό. Και ίσως για τα ζητήματα αυτά στα οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμα συμφωνία στο Συμβούλιο, Είμαστε εδώ πέρα για να σας ακούσουμε πάρα πολύ προσεκτικά και να λάβουμε υπόψη τα σχόλιά σας. Επίσης ε, θα ήθελα να αναφερθώ σε μια άλλη σημαντική προτεραιότητα της ε, Προεδρίας της Κύπρου όσον αφορά την πολιτική συνοχή, την προώθηση δηλαδή της ε, εδαφικής προσέγγισης. Έχει λοιπόν πλέον η πολιτική συνοχή ένα σημαντικό ρόλο να παίξει για να διαμορφώσει την ε, εδαφική ποικιλομορφία σε κάτι το θετικό. Άρα σκοπεύουμε να να κάνουμε μια σειρά συναντήσεων στην Κύπρο, οι οποίες θα προετοιμάσουν τις συνεδριάσεις των Γενικών Διευθυντών, των Αρμοδίων για την Εδαφική Συνοχή και την Πολιτική Συνοχή και σκοπεύουμε να συνεχίσουμε το έργο των προηγούμενων προεδριών για την πρόθεση και την εφαρμογή της εδαφικής ατζέντα 2020. Επιπλέον η ετήσια ε, σύνοδος των ισιωτικών περιφερειακών περιοχών περιφερειών οι οποίες θα λάβει η χώρα στην Κύπρο θα εστιαστεί ακριβώς στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής στην πολιτική συνοχή τέλος ε, αλλά εξίσου σημαντικό θα διοργανώσουμε ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο των Υπουργών που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχή για να συζητήσουν οι Υπουργοί τον προγραμματισμό για το μέλλον ε, για τα κονδύλια αυτά στο πλαίσιο της νέας μας πολιτικής μας καθώς επίσης και για τον ρόλο της πολιτικής συνοχής για να ε, υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως και η κυρία Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία θα προσκληθούν. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, θα ήθελα και πάλι να εκφράσω την ε, χαρά μου για την παρουσία μου εδώ πέρα σήμερα. Παρουσιάσαμε ένα φιλόδοξο, όπω όλοι το χαρακτηρίσαν, πρόγραμμα για το επόμενο εξάμεινο και θα ήθελα να ζητήσω και πάλι την στήριξή σας. Έχουμε βαρύ πρόγραμμα μπροστά μας, αλλά αναμένω μια επικοδομητική συνεργασία μαζί σας στους επόμενους έξι μήνες, ειδικά στο σημαντικό θέμα της νέας μεταρρύθμισης πολιτικής συνοχής που θα δώσει την δυνατότητα στις περιφερειές μας να επενδύσουν για να βγουν από την κρίση. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να τονίσω πως η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί για να διασφαλίσει πως το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής θα υιοθετηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες συνθήκης και σεβόμενοι τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνοψίζοντας λοιπόν, το Συμβούλιο έχει μία μερική και γενική προσέγγιση και είναι έτοιμο να αρχίσει να συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε να κλείσουμε το στομότερο δυνατόν για να αρχίσουμε να διαθέτουμε κονδύλια το στομότερο δυνατόν το 2014 και βέβαια στοχεύουμε να κλείσει να ολοκληρωθεί το πολιτές μεσονομικό πλαίσιο, όπως είπατε στο στόμο δυνατόν. Κατόπιν, κυρία Πρόεδρε, και εσείς και η αντιπροσωπεία θα προσκληθείτε στην ε, ε, επίσημη συνάντηση για τα θέματα της συνοχής 6 ε, Νοεμβρίου στην Κύπρο και βεβαίω Σεπτέμβριο αναμένουμε και η επίσκεψή σας στην Κύπρο. Υπάρχει, υπάρχουν άλλα ζητήματα στα οποία αναμένουμε την άποψή σας, ζητήματα στα οποία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί κάποια κοινή θέση στο Συμβούλιο και θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προωθήσουμε τις θέσεις του Συμβουλίου και τελειώνω εκφράζοντας την πραγματική μου ευγνωμοσύνη για την γρήγορη και ρεαλιστική προσέγγιση που έχετε οθετήσει στην Επιτροπή σας για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. You, you, you ε, προσπαθήσατε να είστε ρεαλιστικός, αλλά νομίζω πως υπήρχε και μια δόση αισιοδοξία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο πρώτος ο οποίος θα λάβει τον λόγο είναι ο Γιώργος Σταυρακάκης, πρώτος αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, να καλωσορίσω την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου και σας προσωπικά στην Επιτροπή μας και να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι πρόκειται να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης Αναγνωρίζουμε ότι η Κύπρος αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια πολύ κρίσιμη καμπή στις διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής και έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα ενεργήσει, ένας, θα ενεργήσει ως ένας ισχυρός διαμεσολαβητής ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία διαπραγματεύσεις στο τέλος της χρονιάς. Είμαστε σίγουροι ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει κατανοήσει το σημαντικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει η πολιτική συνοχή στην αρχιτεκτονική του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και ότι αποτελεί τον κύριο επενδυτικό εργαλείο που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσκοπεί στην μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την ανάκαμψη, την τόνωση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας και καθώς επίσης τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό το απαιτητικό έργο που έχετε αναλάβει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρο. Πρόεδρε. Ε, <clears throat> κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε. Έχετε αναλάβει ένα πολύ δύσκολο έργο για να φέρετε σε πέρα στη διαπραγμάτευση για πολύ σημαντικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και μεταξύ των διαφόρων καονισμών για να πετύχουμε τους στόχους Ευρώπη 2020 ε, θα έλεγα ότι για μας εδώ ως Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιμείνετε και να καταφέρετε να υπάρχει μια συμφωνία για δεσμευτική συμμετοχή των περιφερειών, των περιφερειακών αρχών στα θέματα της περιφερειακής ανάπτυξης. Δηλαδή θα θέλαμε να μιλήσουμε και να έχουμε στο τέλος αυτής της Προεδρίας πραγματικά μια συμφωνία για την εταιρική σχέση με δεσμευτικό χαρακτήρα, να έχουμε συμβόλαια δηλαδή εταιρικής σχέσης μεταξύ των, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των περιφερειών για τα θέματα της ε, περιφερειακής ανάπτυξης. Η περιφερειακή ανάπτυξη όμως για να είναι ουσιαστική πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή θα πρέπει να ενσωματώνεται στην όλη διαδικασία η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των περιφερειακών αρχών Δηλαδή σχέδια για τις περιφέρειες δεν πρέπει να γίνονται από τα κράτη από μόνα τους, αλλά σε συνεργασία με τις περιφερειακές αρχές, αλλά και με τη συμμετοχή των κοινωνιών σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, πολύ σημαντικό στη διάρκεια της δικιάς σας Προεδρίας είναι να δώσετε όθηση στην πράσινη και κοινωνική καινοτομία και στα θέματα της ε, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή που εκεί κρίνεται και το γεγονός αν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε την καρδιά αλλά και το μυαλό των ανθρώπων για την Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται να εμπνεύσει ξανά τους πολίτες και ένα πραγματικά εργαλείο γι' αυτό είναι να προωθήσει αποτελεσματικά μια πολιτική για την απασχόληση ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Ε, ας μην ξεχνάμε όμως ότι η σημερινή κρίση δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κρίση περιβαλλοντική και κλιματική. Ε, και επειδή εσείς είστε και μια νησιωτική κοινωνία και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει ε, η κλιματική αλλαγή για, για, τις νησιωτικές κοινωνίες και ειδικά για τον νότο της Ευρώπης νομίζω θα πρέπει να δώσετε πολύ μεγάλη έμφαση. Όπως και το θέμα των μακροπεριφερειών. Ο συνάδελφος ο κύριος Αλφονσί θα μιλήσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσετε κι εσείς μια όθηση στην έκθεση Αλφονσί ε, γύρω από αυτά τα θέματα. Και τέλος να τονίσω ότι είναι σημαντικό ότι είστε μια νησιωτική χώρα και άρα θα πρέπει να ενθαρρύνετε και να δώσετε όθηση στα θέματα της νησιωτικότητας. Είτε αυτό αφορά τις συγκοινωνίες, είτε αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος, τα θέματα των μεταφορών ε, ή γενικά τα θέματα της οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βανίστεροι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μιλήσατε και για αισιοδοξία και εσείς. Αυτό έχει μεγάλη σχέση και με την αίσθηση της πραγματικότητας και τη φιλοδοξία που έχει κάποιο σε περίοδους κρίσης και ανασφάλειας να επεξεργάζεται θέματα σε αυτό το επίπεδο. Κυρίως ε, αυτό αισθάνθηκα εγώ και η δική μας Επιτροπή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τα όσα είπατε και τα όσα έχουν προετοιμαστεί από τη Δανική Προεδρία τώρα μπαίνουν σε μια νέα φάση, κάπως διαφορετική. Και έχουμε τώρα μια πρώτη εντολή εμείς για να διασαφήνισουμε κάποια πράγματα. Ε, είπατε και ότι στο Συμβούλιο υπάρχουν κάποια κεφάλαια που προσωρινά έχουν εγκριθεί. Από ό,τι φαίνεται σήμερα και αύριο θα ψηφίσουμε και μετά θα είμαστε και εμείς σε θέση ε, σε αυτό το πακέτο των διαπραγματεύσεων να μπούμε στη συναπόφαση για να διεκπαιρεώσουμε ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα πράγματα. Είναι και δικό μας μέλημα έτσι ώστε ε, να περάσουμε στην οριστική φάση της εξέτασης και ψηφοφορίας. Και χαίρομαι που μας είπατε ότι με ενεργό τρόπο θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Έχετε αυτή την πρόθεση στη ημερήσια διάταξη και πούμε, σε ένα άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο ή και σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων διευθυντών και επίσης ε, απευθύνεται και πρόσκληση να μας δεχτείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ε, την προσωπία μας και οι ε, θα δράξουν αυτή την ευκαιρία. Χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόταση. Και άκουσα και τις φιλοφρονήσεις για τη Δανική Προεδρία. Εσείς μας ενημερώσατε. Ε, αλλά αναζητείται ακόμα, είναι ζητούμενο η ισότητα, η ισοτιμία. Έχουμε ένα νέο ρόλο τώρα ως συνομοθέτες. Και στο παρελθόν τι έγινε και πήγε στραβά. Το Συμβούλιο με κάποια αιμονή ε, προχωρούσε ε, στις διαπραγματεύσεις ε, και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τα λοιπά, που τελικά είναι θέματα συναπόφασης. Γίνεται λόγος για μεταβατικές περιφέρειες, για ένα ταμείο επιδόσεων. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά θα πρέπει να τα συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο επί της ουσίας. Και οπωσδήποτε, γιατί δεν επιτρέπεται με θέματα ε, που είναι ισχύουσα νομοθεσία και ορίζονται και από τη συνδίκη της Λισαβόνας να μην τα σεβόμαστε και να ε, παραβιάζονται και να καταπατώνουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο. Έχουμε κάνει και ερωτήσεις σχετικά και δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Κοινοβούλιο απλώς να συνενεί στο τέλος ή όχι. Εγώ θα ήθελα να το αντιστρέψω. Όχι. Εάν ε, θέλει το Συμβούλιο να διεκπεραιωθούν κάποια πράγματα στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πολύ ωραία, αλλά δώστε και εκεί τη συναπόφαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε παζάρια ε, με κάποια πράγματα που συνειδητά ε, τα έχουμε εντάξει στην νομοθεσία και φαίνεται κάποιο δεν κατάλαβε τότε ότι ήταν ένα πλαίσιο, δεν, όχι μόνο ένα πλαίσιο, αλλά και υποχρεωτικό και δεσμευτικό αυτό. Και τώρα αυτό λαμβάνει σάρκα και οστά. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα οπωσδήποτε θα ε, το συζητήσουμε μαζί και θα ε, το ε, προωθήσουμε. Και ένα τελευταίο. σε θέματα θεομηνιών και φυσικών καταστροφών έχουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης και το Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχει τονίσει ότι θέλει μια πιο ευέλικτη μορφή. Εδώ και χρόνια λέει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπλοκάρει τόσα χρόνια. Και θα ήθελα επιτέλους μια καμπή. Εσείς είστε ε, νησί. Γνωρίζετε πολύ καλά ε, πώς αλλάζουν οι κλιματικές συνθήκες, οι μετρολογικές, πόσα πράγματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα και απρόπτα και θα ήθελα εκεί να προχωρήσετε και αν θέλετε προς τα εκεί θα έχετε την πλήρη υποστήριξή μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ, Κωνσταντσα Κρέλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και ελπίζω να το κάνετε και εσείς τώρα. Όπως είπα, σας άκουσα πολύ προσεκτικά και χαίρομαι για το ότι έχετε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την Προεδρία σας. Η ομάδα μας θα σας ε, στηρίξει στους στόχους σας και χαίρομαι που ακούω πως ε, θέλετε να ολοκληρώσετε το MFF σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ακριβώς εκεί έχω μία ερώτηση γιατί βεβαίως υπέβαλε ένα διαπραγματευτικό κουτί η Δανέζικη Προεδρία όπου είχαμε ένα 80% ζητημάτων στη συναπόφαση για την πολιτική συνοχή και υποθέτω πως θα το λάβει αυτό υπόψη η Προεδρία σας και δεν θα λάβει αποφάσεις για το MFF οι οποίες θα έπρεπε να λαμβάνονται στην ε, συναπόφαση και να μην ε, προκαταλάβει αποφάσεις οι οποίες μετά θα δυσκολέψουν τις ε, διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο. Θέλω να σας αποτρέψω αυτό να κάνετε κάτι τέτοιο. Το έχουμε πει πολλές φορές και στην Προεδρία της Δανίας μας έλεγαν ναι έτσι θα γίνουν τα πράγματα αλλά ανησυχώ πως ε, θα γίνει ίσως κάποια προσπάθεια να εξασθενήσει εδώ πέρα του Κοινοβουλίου και αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία λέτε για την πολιτική συνοχή χαίρομαι για το ότι είμαστε σε μια γραμμή πολιτική συνοχής ε, και Ευρώπη 2020 και αυτά τα δύο είναι θετικά και μπορούν να αποτελέσουν ένα πρόγραμμα επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά εδώ πέρα οι ομιλίες της Προεδρίας είναι πάντα καλά προετοιμασμένες ακούω όπως λέτε πως θέλετε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο ωραία πράγματα αυτά αλλά εμείς θέλουμε περισσότερα η συνθήκη δεν λέει στενή συνεργασία λέει συναπόφαση και Θέλω να το πω αυτό ευθύς εξ αρχής ξεκάθαρα. Ακούσατε πως θα ψηφίσουμε για διαπραγματευτική εντολή με το Συμβούλιο ε, αργότερα. Το παίρνουμε σοβαρά αυτό το πράγμα. Πρέπει και εσείς να διαπραγματευτείτε μαζί μας. Και ελπίζω να λάβετε υπόψη στις διαπραγματεύσεις σας πως ε, χρειάζεται αρκετή ευελιξία για διαπραγματεύσεις. Αλλιώς είναι τα πράγματα δύσκολα. Θεωρώ μεγάλους στόχους ε, τους οποίους περιγράψατε, συμφωνούμε. Θέλουμε μια σύγχρονη πολιτική συνοχή που βασίζεται στην αλληλεγγύη, αλλά ε, επίσης ε, στοχεύει σε αποτελέσματα, στοχεύει ε, στο να ενισχύσει τις ασθενέστερες περιφέρειες των κρατών μελών να προχωρήσουν, να εφαρμόσουν τους κοινούς μας στόχους. Οπωσδήποτε υπάρχουν ε, πολλοί τομείς ε, στους οποίους έχουμε και διαφορετικές ε, προσεγγίσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ελπίζω το συντομότερο δυνατόν να μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντς. Νομίζω μπορούμε να ζητήσουμε από τον κύριο Υπουργό να απαντήσει στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όσους μίλησαν. Θα ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο για το αρχικό δικό σας σχόλιο και το σχόλιο του κυρίου Φανινής για την αισιοδοξία. Ξέρετε, προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι και φιλόδοξοι, αλλά με τρόπο ρεαλιστικό. Και ταπεινό. Σεμνό και ταπεινό θα έλεγα. Έχουμε όμως και αποφασιστικότητα για να, έχουμε, για να επιτύχουμε αποτελέσματα. Δεν θέλουμε απλά να κάνουμε το καθήκον μας. Αν θέλετε, θέλουμε να προχωρήσουμε και λίγο παραπέρα. Με σεβασμό σε όλους τους εμπλεκομένους και ως άτομα και ως θεσμικά όργανα. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας για τη συνεργασία. Τον κύριο Σταυρακάκη για τα καλά του λόγια και τον κύριο Χρυσόγελο επίσης για τα καλά του λόγια και για ε, τα θέματα τα οποία έχει γύρει. Ε, αναφέρθηκε κυρίως στην συμφωνία για την ε, δεσμευτική συμμετοχή των περιφερειών. Υπάρχουν κάποια στοιχεία για την, την, την εταιρικότητα γενικά που είναι, υπάρχουν ήδη στην, στην, στους κανονισμούς. Ε, εμείς είμαστε έτοιμοι να τα συζητήσουμε όχι μόνο για τη συμμετοχή των περιφερειών αλλά και των άλλων εταίρων, ίσως κοινωνικών εταίρων και άλλων εταίρων που μπορεί ε, να τους ε, αφορά το, το ζήτημα αυτό. θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα αλλά βεβαίως σημειώνουμε, σημειώνουμε αυτά που μας είπατε και ό,τι μας αφορά δεν έχουμε κανένα απολύτως λόγο. Αντίθετα νομίζουμε ότι η ιδέα είναι πάρα πολύ καλή. Πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό και στα πλαίσια του Συμβουλίου και σε σχέση με το τι ε, θέλουν και τα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα και το τι θα ακούσουμε από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό του. Ε, για την ε, περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή, για την κλιματική αλλαγή δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, και βεβαίως έχουμε σημειώσει αυτά που μας είπατε για τις μακροπεριφέρειες, για την έκθεση αλφονσή και θα λάβουμε απολύτω υπόψη ε, τα όσα θα περιέχονται στην έκθεση αυτή. Το ίδιο ισχύει βεβαίω για την νησιωτικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε εμεί σε αυτό το ζήτημα. Έχει να κάνει με την ε, γεωγραφική διάσταση στην οποία αναφερθήκαμε, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και στι ε, ιδιαιτερότητε των, των νήσων γενικότερα και νησιωτικών κρατών επιπλέον. Έχουμε και όλες τι ιστορίε με ε, ultra-peripheral ε, regions και ούτω καθεξής είναι ζητήματα πολύ σημαντικά, πολύ σοβαρά για μας και τα οποία θα λάβουμε πλήρως υπόψη. Ε, on Mr. Nistelrooy's comment on co-decision, and this was also raised by Madam Krell, yes, indeed, I understand. Ναι, κυρία Κρέλ, κατανοώ ότι το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει κάποια συνένεση. Ε, ε, στο διαπραγματευτικό κουτί θα μπουν και κάποια θέματα συναπόφασης θέλετε εσείς. Αλλά αυτά ε, είναι για να βοηθήσουν τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Σε καμία περίπτωση δεν προεξοφλούν ότι θα ληφθεί οδήποτε απόφαση από αυτόν χωρίς να γίνει σεβαστή διαδικασία συναπόφασης. Μπορείτε να το εκλάβετε αν θέλετε σας παρακαλώ ως εσωτερική κουζίνα του Συμβουλίου είναι δικά μα θέματα, αυτά εσωτερικά, δεν χρειάζεται να τα γνωρίζετε. Εάν έρθω ποτέ και σας πω ότι αυτό είναι δεχτείτε το ή όχι ή απορρίψτε το, ε, μπορείτε να με... και να με διαολοστείλετε, αν θέλετε να το πω έτσι. Ε, και η Δανική Προεδρία... Ε, προσπάθησε να διασκεδάσει κάποιες ανησυχίες λέγοντας ότι απλώς ε, εστιάζουμε, εντοπίζουμε κάποια σημεία, ε, τα επισημαίνουμε χωρίς να χρειαστεί ε, να ακολουθήσουμε την τυπική, σωστή διαδικασία. Βεβαίως και σεβόμαστε το θεσμικό πλαίσιο και τη συναπόφαση και τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα προνόμια του. Ο κύριος Ρόι αναφέρθηκε στο Ταμείο Λεγγύης και το εξετάζουμε αυτό το καιρό, τη δομή και την ευελιξία που μπορούμε να το διασφαλίσουμε. Με μεγάλη χαρά να το συζητήσουμε περαιτέρω μαζί σας και να λάβουμε υπόψη κάποια ζητήματα ε, που θα διαβιβάσουμε στο Συμβούλιο και θα ε, φροντίσουμε όσο μπορούμε να καλύψουμε ε, την προσέγγιση αυτή και να επιτύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση. Και τέλος, χωρίς να είναι αυτό το λιγότερο σημαντικό, θα ήθελα να πω ότι, εξ γνωρίζω, αύριο η ομάδα μας συνεδριάζει με ε, την Πρόεδρο και τους συζητητές για να βγούμε σε ένα διάλογο διμερή, τριμερή, όπως θέλετε πείτε το άτυπο, μη διάλογο, γιατί ακόμα δεν έχουμε γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο. είναι μερικές ακόμα οι... Ε, άρα, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, έτσι θα είναι και μερική τριμερής διάλογη, όχι συνολική. Εν πάση περιπτώσει, θα έρθουμε σε επαφή, θα συζητήσουμε και θα προσπαθούμε να ε, τα δούμε εκ του και θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό για να προχωρήσουμε και για να επιτύχουμε πρόοδο στα στοιχεία όπου δεν είναι ακόμα ολική, μερική είναι η θέση του Συμβουλίου, αλλά και κάπου που δεν έχουμε ακόμα καταλήξει θα είναι πολύ χρήσιμο ε, και θα μας βοηθήσει να ακούσουμε τη δική σας άποψη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, αναλαμβάνετε την Προεδρία της Ένωσης μετά από τη Δανία, την Ουγγαρία, την Πολωνία Οπότε εγώ ως νησιώτης ε, Κορσικανός ε, σας χαιρετίζω όλος ιδιαιτέρως. Είμαι πολύ ε, ευτυχής που βλέπουμε πάλι μια προεδρία μεσογειακή με, νέα, με άλλου είδους οπτική για την Ευρώπη. Ξέρουμε πολύ καλά πόσες δυσκολίες διανύει ο μεσογειακός χώρος και θέλω να ξέρω αν η Κυπριακή Προεδρία σκοπεύει να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για τον μεσογειακό χώρο έχετε δεσμευτεί να, να δώσετε συνέχεια στην έκθεση που έχει ψηφίσει το Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μετά από δική μου πρόταση γιατί πιστεύω πως είναι σημαντικό να δοθεί ένα μήνυμα ελπίδας και ένα μήνυμα για το μέλλον ε, ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση την τόσο τεταμένη και δύσκολη και από πλευρές κοινή γνώμης, όχι μόνο από άποψη λογαριασμών, εθνικών λογαριασμών. Ο κύριος Βλάσακ. E, Ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και στο παρελθόν, κυρία Κρέλ, κύριε Φανίστελβοη, δηλαδή συγκεκριμένα το νομικό πλαίσιο. Γνωρίζουμε όλοι πως ε, στο τέλος θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και το ερώτημά μου είναι το εξής. Θεωρείτε πως ε, θα μας ε, ενημερώνετε διαρκώς για τις διαβουλεύσεις εντός του Συμβουλίου. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά την πολιτική συνοχή. Όπως ξέρετε, δεν ε, συμφωνούμε πλήρως για ε, ένα ποσό γύρω στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ για το μέσο συνδέοντας ε, την Ευρώπη. υπάρχει κάποιο περιθώριο συμβιβασμού εδώ πέρα και το τρίτο μου ερώτημα αφορά τον ΦΠΑ και ε, πρέπει να γνωρίσουμε πως εάν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ε, ΦΠΑ ως ε, επιλέξιμη δαπάνη ή θα γίνει πάρα πολύ δύσκολη θέση πολλών κρατών μελών. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Σκουσμάνης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να τονίσω κάτι για τον προπολογισμό του επομένου έτους ε, και ούτε καν για το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Κύριε Πρόεδρε, ο τριμερής διάλογος μεταξύ Συμβουλίου Κοινοβουλίου και Κομισιόν κατέληξε σε πλήρη διαφωνία. Ξέρετε πως η Κομισιόν ε, κατέθεσε μία πρόταση αύξηση των πληρωμών για τα επόμενα χρόνια κατά 6,8%. Μεγάλο ποσοστό, αλλά αν δείτε τα διάθετα κονδύλια Πρέπει γι' αυτό να αντιπαλέψουμε αυτά τα 210 δισεκατομμύρια ευρώ. Η απάντηση του Συμβουλίου ήταν να από το 6,8 να πάει στο κάτω από το 2%. Δεν υπήρξε εξήγηση γιατί κυρίως βεβαίω συμμετείχαν οι πρέσβεις της Κορεπέρα, όχι οι υπουργοί, αλλά το πρόβλημα είναι πως εάν επιμείνει σε αυτή τη θέση το Συμβούλιο, τα αδιάστα θα αυξηθούν κατά 17 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Με απλά λόγια σημαίνει πως εάν περάσει τη θέση του το Συμβούλιο και ελαχιστοποιήσει την αύξηση πληρωμών σε λιγότερο από 2% τα λεφτά κατόπιν θα αναβληθούν και θα πάνε στο επόμενο πολιτισμό μεσονομικό πλαίσιο 2014-2020 και τόσο μεγάλο ποσό το οποίο νομικά πρέπει να εκταμιευτεί γιατί ξέρετε πως αυτό το οποίο επιτρέπεται στο Ταμείο Συνοχής ε, για τις χώρες που είναι κάτω από το 85% ε, του ΑΕΠ κατά κεφαλή είναι το 2017. Και δεν είναι πλέον ε, μετά δυνατόν να εκταμιευθούν αυτά τα λεφτά. Οπότε, αν προσπαθήσει το Συμβούλιο να εξοικονομήσει λεφτά, από ό,τι φαίνεται, το τελευταίο έτος το οποίο θα ολοκληρωθεί με πληρωμές θα επιδεινώσει το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και όλους τους στόχους μας και τα όνειρά μας ε, κτλ. Οπότε Παρακαλώ να δώσετε ιδιαίτερο βάρο στον προκλήσιμο του επόμενου έτου 2013 γιατί το 65% των αδιαθέτων είναι κονδύλια τη συνοχή και σημαντικό είναι να ολοκληρώσουμε ό,τι μπορούμε να ολοκληρώσουμε στο τέλος αυτή τη 7 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Σαγκουράκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είναι γεγονό ότι αναλαμβάνετε μια μεγάλη καυτή πατάτα ε, και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη διαχείριση του προβλήματος. Ε, νομίζω σε εσά ιδιαίτερα είναι ιδιαίτερα καθαρό ότι όταν μιλάμε για καυτή πατάτα εννοούμε κυρίως το ζήτημα ότι έχετε αναλάβει ένα έργο σε μια εποχή που οξύνεται η καπιταλιστική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ιδιαίτερη ιδιομορφία ε, του προβλήματος για σας είναι ότι πρέπει να κλείσετε μια σειρά από χρηματοπιστωτικά ζητήματα, ζητήματα επενδύσεων, το PDP και το θέμα των Ευρωπαϊκών Ταμείων, σε μια εποχή που είναι τελείως αβέβαιον το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η μεγάλη πατάτα για την Κυπριακή ε, Δημοκρατία. Ε, θα έχετε υπόψη σας φυσικά ότι η Ελλάδα και άλλες δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε προγράμματα συγκεκριμένα λόγω της καπιταλιστικής κρίσης. Καροδοκούν ε, μνημόνια για την Ισπανία και για την ε, Ιταλία στα πλαίσια των τελευταίων αποφάσεων και της Συνόδου Κορυφής και γενικώ η κρίση θα οξυνθεί και θα συμπεριλάβει και τις μεγαλύτερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα οι προοπτικές είναι πάρα πολύ δύσκολες, δυσιόνιες. Η επίθεση στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους θα οξυνθεί ακόμα περισσότερο και τα αδιέξοδα που μας έχουν οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους, τους τομείς της συνοχής ε, οι λεγόμενοι θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο. Εγώ έχω δύο παρατηρήσεις να κάνω κύριε Υπουργέ και θα ήθελα την θέση σας. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι κατά την άποψή μας στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολιτική συνοχής και εξηγούμε. Δεν θα μπορούσε εξάλλου να υπάρχει γιατί η, η, βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο καπιταλιστικών χωρών, υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός, υπάρχει η λεγόμενη ανισόμετρη ανάπτυξη. Όμως με την και με την ένταξη εξ ολοκλήρου των πολιτικών συνοχής στους στόχους της Ευρώπης 2020 Συνοχή δεν υπάρχει ούτε καν στα λόγια από εδώ και στο εξή. Και αυτό γιατί μια ενιαία πολιτική του, του είδους ε, Ευρώπη 2020 όπως και προηγούμενα οι πολιτικές της, ε, στα πλαίσια της Λισαβόνας ή αν θέλετε στα πλαίσια και της ενισχυμένης οικονομικής διαχείρισης βεβαίως οδηγούν σε απόκληση ε, τις, αδύνατες, πιο αδύνατες χώρες μέλη και είναι ακριβώς το πρόβλημα που έχουμε με τον νότο της Ευρώπης. Άρα η εφαρμογή μιας παρόμοιας πολιτικής όπως είναι η Ευρώπη 2020 χωρίς καν να παίρνετε υπόψη ότι θα υπάρχει απόκληση θα οξύνει ακόμα περισσότερο το πρόβλημα. Και βεβαίως θα οξύνει το πρόβλημα προς όφελος του μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου, ευρωπαϊκού και ντόπιου. Δεύτερο ζήτημα που ήθελα την άποψή σας είναι το εξής. Πρόσφατα αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορφής στις 28 Ιουνίου το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη ύψους 120 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τα 55 δις είναι επιστροφές, όπως υπόθηκε ε, επισήμως, από μία απορροφημένα ταμεία του, ε, ε, μια απορροφημένους πόρους του ταμείου, του ταμείου Συνοχής, των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Θα συνεχιστεί αυτή, αυτό το βιολί και στο μέλλον, έχετε υπόψη σας. Δεν θέλω να, να, χρεώσω στην Κυπριακή Δημοκρατία όλες τις πληγές του Φαραώ. Όμως αυτό το πράγμα θα το έχουμε και μελλοντικά ποια θα είναι η σχέση του, του, Σύμφωνου Ανάπτυξης με, ε, τα προγράμματα ε, του, Ταμείου Συνοχής. Και κυρίως εμεί εμείς διαφωνούμε κάθετα με το να χρησιμοποιούνται τα χρήματα αυτά και του Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής με έργα που δεν έχουν καμία σχέση με τις αναπτυξιακές ανάγκες των χωρών. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα έχουμε 30 κλάδους που μπορούν να προωθήσουν μια ανάπτυξη προς όφελο των εργαζομένων και τη χώρα. και από αυτούς μόνο τρεις κλάδοι είναι στου στόχου τη Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much. And the last speaker is... Uh, ευχαριστώ. Έρικα Μάνερ θα ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό, με χαρά σας άκουσα και βλέπω πως ε, έχετε μεγάλο ενθουσιασμό για τους επόμενους έξι μήνες και για την πολιτική συνοχή. Ε, βεβαίως θα είναι δύσκολη αυτοί οι έξι μήνες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Όπως ε, είπαν ήδη πολλοί ομιλητές, είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα γιατί θα πρέπει να επιτύχουμε συμφωνίες φέτος και για την πολιτική συνοχής για να μπορέσουν και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τα προγραμματά τους όσον αφορά τώρα το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ιδιαίτερα θετικό το ότι υπερασπίζεστε την ε, πολιτική συνοχής και θα ήθελα να μάθω ποια θα είναι η πολιτική σας όταν θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε εντός αγωγικών για την περιφερειακή πολιτική και τη γεωργική πολιτική γιατί βεβαίως ε, αυτές είναι μεγάλες πολιτικές και απορροφούν τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού και είναι θετικό το ότι τονίσατε ε, τις ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις, νησιωτικές περιοχές, ε, θαλάσσιες περιοχές και λοιπές απομακρυσμένες περιφέρειες. Πρέπει να δείτε και τις ιδιαίτερα αρεοκατοικημένες περιφέρειες που έχουν δική τους γραμμή του προϋπολογισμού και αν θέλουμε να τις προωθήσουμε πρέπει να διασφαλίσουμε τουλάχιστον τα 926 εκατομμύρια ευρώ που αντιστοιχούν σε αυτές γιατί είναι σημαντικό για εμάς να παραπίνουν οι πληρωμές στο ε, επίπεδο που είναι αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το πρόγραμμα για την εδαφική συνεργασία. Είμαι εισηγήτρια εγώ για αυτό το θέμα και θα ήθελα άρα να δραστηριοποιηθείτε σε αυτόν τον τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορούμε τώρα να κλείσουμε το κατάλογο των ε, μελών της Επίτροπης. Μίλησαν. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Αυτή ήταν η τελευταία ομιλήτρια. Θα ήθελα να παρακαλέσω και πάλι τον κύριο Υπουργό να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, για να απαντήσω στο ερώτημα του κυρίου Αλφονσί. Βεβαίως αποδίδουμε μια ιδιαίτερη σημασία στη θάλασσά μας, στη Μεσόγειό μας. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ακριβώς για να εστιάσουμε στη μεσογειακή πολιτική. Γνωρίζετε ότι είναι και στοιχείο των προτεραιοτήτων μας πολιτική γειτονίας προς νότο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργαζόμαστε πάρα πολύ προς την κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα σύνδεσης της ε, δράσης της εκπεριτροπής ε, προεδρίας και της υπάτης εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δηλαδή, στα πλαίσια των δικών μας αρμοδιοτήτων θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία γνωρίζετε ότι αυτή η συνεργασία ανέκαθεν ήταν προβληματική. 13 ε, έτη αναλώσαμε ε, στην μεσογειακή πολιτική που στην καλύτερη περίπτωση ε, απορροφήθηκαν 25% των κονδυλίων που είχαν δεσμευτεί. Ακολούθησε η Ένωση για τη Μεσόγειο, η οποία ουδέποτε απογειώθηκε, να το πω έτσι, για διάφορους πολιτικούς λόγους. Και πέρα από τις πολιτικές δηλώσεις, τώρα όπως είπατε και εσείς θα πρέπει να δουλέψουμε επί τόπου. Δεν είναι θέμα χρημάτων ούτε μέσων. Είναι ζήτημα ε, βούλησης. Μπορούμε σε όλες αυτές τις χώρες να βρούμε ε, μικρές ε, ομάδες ε, πληθυσμού και να εργαστούμε μαζί τους όχι για αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά για να τους συνοδεύσουμε στη μετάβασή τους προς τη δημοκρατία. Και αυτό θα είναι πραγματική ε, λοιπόν στη συνέχεια εδραίωση αυτής της διακασίας ε, εκδημοκρατισμού και ε, θα ανταποκροθεί και στις προσδοκίες των λαών, να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται κάποια πράγματα. Γιατί έχουμε τον εξή φόβο, ότι αυτά που παρατηρούμε τώρα στην περιοχή αυτή, να είναι για κάποιες πολιτικές δυνάμεις μια ευκαιρία χειραγώγησης της διαδικασίας εκδημοκρατισμού για να ε, συνεχίσουν να ε, επιδιώκουν άλλου είδους στόχους. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε κάποια ε, ολοκληρωτικά ή αυταρχικά καθεστώτα από κάποια άλλα αυταρχικά καθεστώτα. Θα πρέπει να βρούμε διάβλους επικοινωνίας, πολλούς, και να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε πρόσβαση σε αυτή την κοινωνία με πολυφωνία. Και είτε πρόκειται για πολίτες, για μη κυβερνητικέ οργανώσεις, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις αυτών των κρατών, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάπου υπάρχουν δυνατότητες άμεσης εταιρική σχέσης και συνεργασίας με ε, δυνάμεις στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε έτσι θα συσφίξουμε τους δεσμούς μας για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και ε, πολυφωνικές κοινωνίες και κοινωνίες όπου η αρχή που έχουμε για τη συνεργασία μας more for more, περισσότερα για περισσότερο, θα λάβουν και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δηλαδή, για να επιτύχουμε περισσότερα σε επίπεδο κυβερνήσεων και κρατών, εμ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να επιτρέψουν Ε, την επαφή και τη συνεργασία σε επίπεδο κατώτερο του επίσημου κρατικού και κυβερνητικού. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν κονδύλια τα οποία έχουν δεσμευτεί για αυτές τις πολιτικές, ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης διαθέτουν τέτοια κονδύλια και θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε ε, τον τρόπο για να συνεργαστούμε πιο αποτελεσματικά. Για αυτή τη συνεργασία που όπως σας είπα είναι πραγματικά ιδιαίτερα προσφυλής μας και έχουμε και εμείς ιδιαίτερη ευαισθησία για αυτή. Ταυτόχρονα όμως η Μεσόγειος έχει και ιδιαιτερότητες που μας αφορούν όλους μας. Ε, όχι μόνο η Νότια Όχθη, Κορσική, Κύπρος, Κρήτη, όλα τα νησιά μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι και ε, στην εργασία μας στην εδαφική συνοχή να βρούμε τον τρόπο να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι ιδιαιτερότητες θα ε, ληφθούν υπόψη. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο κύριος Βλάσακ. Είναι γεγονός ότι ε, θα προσπαθήσουμε να ε, τηρούμε πάντα ενήμερο το κοινοβούλιο όσο μπορούμε. Έχουμε ε, αυτό το modus operandi με συνεδριάσεις πριν και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Αν χρειαζόμαστε όμως έκτακτες ειδικέ ανταλλαγές απόψεων, είμαστε στη διάθεσή σας. και με άτυπο τρόπο να έχουμε ενημέρωση και διάλογο με το Κοινοβούλιο. Έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να είναι πλήρως ενήμερο για την κατάσταση των πραγμάτων και την πρόοδο των εργασιών στο Συμβούλιο για διάφορα θέματα. Είτε πρόκειται για τα θέματα συνοχής που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή σας, αλλά είτε και αν πρόκειται ε, για τις γενικές εξελίξεις, για το PDP, διότι γνωρίζετε ότι συνδέονται άμεσα. Για τα 10 δισεκατομμύρια που έχουν προσημειωθεί στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη, τη διευκόλυνση αυτή ότι θα προέλθουν από τη συνοχή. Εγώ δεν μπορώ να λάβω θέση εκεί. δίστανται οι απόψεις μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να το χειριστούμε, διότι εμένα το πρόβλημά μου ποιο είναι ως Προεδρία. δεν είναι μόνο τα 10, είναι και 15, γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη ε, που θέλουν να το μειώσουν 20-15 κάθε χώρο. Αν είναι 50 λοιπόν, 20, 15, 25 θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα πιάσουν τόπο τα χρήματα αυτά. Και για τις μεταφορές, και για την ενέργεια, και για τις τηλεπικοινωνίες. Και βεβαίω, γνωρίζουμε και το θέμα του φόρου τη προστιθέμενης αξίας και εκεί επιμένουν πολλά κράτη-μέλη. Θέλουν να λαμβάνεται υπόψη και να συνυπολογίζεται ο ΦΠΑ. Γνωρίζουμε ότι και το κατανοούμε, είναι θεμητό αυτό ως μέλημα, αλλά και πάλι θα πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό σε επίπεδο ένωσης. Και βεβαίως και το μήνυμά σα θα ληφθεί υπόψη και θα διαβεβαστεί αρμοδίω στο Συμβούλιο. Κύριε Γκοντμάνη. Έχουμε πλήρη επίγνωση ε, του προβλήματος των αδιαθέτων ποσών, των ραλ. και προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα ως πολιτικό ζήτημα και κάποια στιγμή τελικά να το καταστήσουμε τεχνικό. Διότι σήμερα ε, ε ισχύει αυτό που λέτε πολίτος. Έχει καταστεί γνήσιο πολιτικό ζήτημα στις συζητήσεις αυτό. Να δούμε πώς ε, θα το διεκπαιρεώσουμε και ξέρουμε ότι τα περισσότερα διάθετα κονδύλια είναι κονδύλια της συνοχής. Θα πρέπει να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα ε, της πολιτικής συνοχής και την αποδοτικότητα τη δική μας. Αυτό είναι του μέλλοντος. Για τον προπολογισμό του 2013 ομολογώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα, διότι υπάρχει βέβαια αυτή η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 6, κάτι αύξηση ε, στις πιστώσεις πληρωμών. Ίσως ε, τρομάξαμε και κάποια κράτη-μέλη που ήθελαν πλήρες πάγωμα του προϋπολογισμού. Δηλαδή η ε, Προεδρία πρέπει τώρα να πλέψει σε πολύ βαθιά νερά. Δεν ξέρω εάν υπερβαίνω την εντολή μου και σας αποκαλύπτω κανένα μυστικό, αλλά υπάρχει ένα είδος συμφωνίας στο Συμβούλιο, θέλετε λέτε, ενισχυμένη πλειοψηφία για αύξηση ε, κατά 2,79 είναι λιγότερο από εκείνο που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περισσότερο από εκείνο που εσείς ε, φοβηθήκατε και εμείς φοβηθήκαμε, ότι είναι κάτω από 2%. Για να δούμε αν θα ισχύσει, θα παραμείνει έτσι αυτή η συμφωνία και αν θα μπορέσει να αποτελέσει βάση για τη συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. I to... Έρχομαι τώρα στα ελληνικά. Ε, κύριε Αγκουράκη, έχετε δίκιο ότι έχουμε καυτές πατάτες και σε μια σειρά από θέματα και ξέρετε η δική μας φιλοσοφία στο τέλος της ημέρας είναι ε, όταν έχει κανείς ε, καυτές πατάτες και τέτοια δύσκολα θέματα δεν μπορεί να περιμένει να λυθούν από μόνο τους τα προβλήματα. Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης τους είναι να ανασκουμποθείς, να σηκώσει τα μανίκια και να αρχίσεις να δουλεύεις και στην πράξη να αλλάξει τα δεδομένα για να μπορέσει να, κάνεις, να φέρεις αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε. Είναι σίγουρο ότι σε μερικά ζητήματα ίσως να προχωρούμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα αλλά ε, πρέπει, πρέπει να κάνουμε κάτι πρέπει να εργαστούμε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε βήμα με βήμα ε, δεν, δεν πιστεύω ότι έχουμε μαγικές λύσεις να προτείνουμε το μόνο που έχουμε στη διάθεσή μας είναι ε, την ευαισθησία την κοινωνική ευαισθησία που απαιτείται και τη βούληση να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ξέρετε, υπάρχουν στη στρατηγική αυτή και κάποιοι απόλυτα μετρήσιμοι στόχοι που αν επιτευχθούν σίγουρα θα συμβάλλουν στην βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης της Ευρώπης. Ε, και παραδείγματος χάρη ξέρετε ότι υπάρχει η ιδέα ότι πρέπει ε, να έχουμε τουλάχιστον 75% του ενεργού πληθυσμού που να έχει απασχόληση υπάρχει αυτή, ο στόχος του να έχουμε 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος να πηγαίνει στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Έχουμε τους ε, περιβαλλοντικούς στόχους ε, της Ευρώπης Έχουμε τον, ε, το θέμα του αναλφαβητισμού. Έχουμε διάφορους μετρήσιμους και συγκεκριμένους στόχους που αν επιτευχθούν πιστεύω ότι θα είναι σημαντικοί για την Ένωση και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αν θέλετε για να δώσουμε ένα πιο κοινωνικό πρόσωπο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη φέρουμε τελικά πιο κοντά στους πολίτες και βεβαίως και τους πολίτες στο μέτρο του δυνατού ε, πιο κοντά στην Ένωση. On ε, Mrs. Manner's question, σε σχέση με την ερώτηση της κυρίας Μάνερ, όπως είπα προηγουμένως, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής και βεβαίως επιθυμούμε η πολιτική αυτή να έχει πραγματική προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μόνες αλλαγές που προβλέπουμε είναι και είναι κοινή μας φιλοδοξία αυτό να έχουμε ένα πιο εξυγχρονισμένο και αποτελεσματικό είδος πολιτικής που να είναι πιο ολοκληρωμένη και να λαμβάνει υπόψη και τα διαμεθοριακά ζητήματα και όλα αυτά τα θέματα που τελικά θα επιτρέψουν να υπάρχει μεγαλύτερη συνέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την οικονομία κλίμακας στις δαπάνες μας για να είμαστε και αποδοτικοί και αποτελεσματικοί και αηφόροι και ταυτόχρονα βέβαιοι και να πείσουμε και τους λαούς μας και κάποιες κυβερνήσεις που είναι άκρος ε, επιφυλακτικές ότι κάθε ευρώ που δαπανούμε πιάνει τόπο. Και αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και να το αισθάνονται με αυτόν τον τρόπο και να το εκλαμβάνουν έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν φανταστική αυτή η ανταλλαγή απόψεων, εξαιρετικά χρήσιμη για μας και προσβλέπουμε σε συνεργασία μαζί σας. Ευχαριστώ. Και συνέχιση αυτής. Thank you, Minister. Uh, very much. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Dear colleagues. Συνάδελφοι, συνεδριάζει η Επιτροπή. Σας παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, σε ονόματος όλων σας διαβεβαιώ πως ε, και η Επιτροπή μας θα εργαστεί σκληρά τους επόμενους μήνες και η φιλοδοξία μας είναι επίσης ρεαλιστική, αλλά ελπίζω οι φιλοδοξίες αυτές να μας οδηγήσουν σε επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και για το ΠΟΔΟΠΟΥ και το νομοθετικό πλαίσιο. Ε, εκτιμούμε βεβαίως και την συνεργασία που είχαμε με τους δικούς σας ε, συνεργάτες ε, και βεβαίως θα θέλαμε στο τέλος της Προεδρίας να έρθετε και να μας πείτε πως η αποστολή εξετελέστη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, um, uh, Είναι δέκα και μισή ήδη αγαπητοί συνάδελφοι, οπότε νομίζω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις δύο ψηφοφορίες πριν περάσουμε στον κανονισμό στο σημείο 7 λοιπόν αλλά πρώτα απ' όλα να ελέγξουμε τα μηχανήματα παρακαλώ βάλτε λοιπόν τις κάρτες σας στο μηχάνημα άρχιτη ψηφοφορία ε, Dear colleagues, we have 41 41 κάρτες είναι στο μηχάνημα και μόνο 30 συνάδελφοι ψηφίζουν. Για κοιτάξτε το. Mm, κάποιοι είναι παραπάνω από τους σοσιαλιστές, γι' αυτό παρακαλώ να ψηφίσετε όλοι. Τέσσερις ακόμη δεν έχουν ψηφίσει. Σας ελέγχουμε, τα βλέπει τα πάντα ο μεγάλος αδερφός οι τέσσερις κάρτες δεν λειτουργούν ή δεν είναι εδώ πέρα συνάδελφοι. 42 κάρτες είναι στο μηχάνημα και μόνο 38 ψηφίζουν. Και πάλι παραπάνω είναι από τους σοσιαλιστές. Ένας παραπάνω. So what we need Τρία άτομα πρέπει να ελέγξουν τις κάρτες τους γιατί υπάρχει ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Και ε, ακόμα ένας σοσιαλιστής παραπάνω. Μπορεί κάποιος σοσιαλιστής να βγάλει την κάρτα του που είναι υπεράριθμος. Substitute less. It's Ένας αναπληρωτής λιγότερος, ωραία, εντάξει, και κάποιος δεν ψήφισε. Λοιπόν, ξεκινάμε το σημείο 7, έκθεση στη Τυρολιάνου. Τροπολογία 36 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. συμβιβαστική 2, όχι. Ψηφίζουμε όλα αυτά. So, amendment 11. Τροπολογία 11, 38, 39, 40, 41, 42 ταυτόσιμες υπέρ κατά συνάδελφοι ε, να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία τις πέντε αυτές ταυτόσιμες τροπολογίες πέρας 21 με 21 ισοψηφία απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 13 υπέρ κατά νομίζω πως έχει απορριφθεί αλλά να, να επαληθεύσουμε γρήγορα γιατί δεν είναι σαφές πέρας Απορρίπτεται. Τροπολογία 13, 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ. Κατά αποχές. Τσίμα τσίμα μου φαίνεται να την επαληθεύσουμε. Πέρασε. απορρίπτεται μεγάλη διαφορά περνάμε στην 15 υπέρ υπέρ κατά εποχές δεκτή 16 υπέρ κατά εποχές δεκτή 17 υπέρ κατά εποχές δεκτή 18 υπέρ κατά δεν μπορώ να διακρίνω να το επαληθεύσουμε πέρας απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε τη 47 πέρας δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορριπτούνται 50 κατά 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ να υποληθεύσουμε την 52 πέρας Δεκτή. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν, ξε, δεν ξέρω. Να επαληθεύσουμε την 53. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Νομίζω πως η ίδια πλειοψηφία είναι να επαληθεύσουμε όμως και την 54 γιατί δεν μπορώ να κρίνω. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτεί. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριπτεί. 58 υπέρ να επαληθεύσουμε την 57 πέρας δεκτή ε, α με συγχωρείτε απορρίπτεται ναι ναι έχετε δίκιο 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε Άρχεται η ψηφοφορία. Δεκτή. 62 υπέρ κατά εποχές. Να, να υπολυθεύσουμε. Άρχιε ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. Η 22 ήταν συμβατή. Οπότε δεν την ψηφίζουμε. Να την ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά από αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε την 68 άρχιτη ψηφοφορία πέρας δεκτή συνάδελφοι όταν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά έτσι να είστε λίγο γρήγοροι Είσαι, δεν ξέρω, είστε το μηχάνημα 69 υπέρ κατά ναι, δεν μπορώ να διακρίνω. Να επαληθεύσουμε την 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. Ε, 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριφθείτε. Εκτιμώντα συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε. Συμβαστική 4. Ναι, δεν μπορεί να κλείσει ψηφοφορία γιατί δεν ψηφίζει ο κόσμος. Πέρασε εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία... Ναι. 27. Ποιος είναι υπέρ? Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε. Πέρας και έχει απορριφθεί. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 6 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε την 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχη ψηφοφορία Συγχαρητήρια. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Και στην Ευρωπαϊκές Δημογραφικές Στατιστικές. Can we start the vote? Amendment 11, who's in favor? Μπορούμε να αρχίσουμε. Η τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ 14, συγγνώμη, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 6, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Η 7, χωριστή ψηφοφορία, ε, τμήμα πρώτο υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 1, είναι σε σκέψη υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 8 δεν ψηφίζεται. Ψηφίζετε, ωραία, ψηφίζουμε 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα. Αποτέλεσμα 42 υπέρ, 4 αποχές. Μπράβο σας και συγχαρητήρια. Τώρα αγαπητοί συνάδελφοι μάλλον πρέπει να ρωτήσω αν θέλετε να βγείτε να πάτε τουαλέτα ή τίποτα τέτοιο γιατί έχουμε μαραθώνια ψηφοφορία. Και σας ζητώ την υπομονή σας να με ακούσετε λίγο, 3-4 λεπτά, να σας εξηγήσω πάρα πολύ καλά κάποια πράγματα. Τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αλλά για να καταλάβουμε όλοι ότι έχουμε ε, την ίδια διαδικασία. Πρέπει να σας πω ότι αποφύσαμε ως Επιτροπή βάσει των συστάσεων που ήρθαν από την ομάδα εργασίας της 26 Απριλίου να ψηφίσουμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας ε, του Ιουλίου για να δοθεί εντολή και να υπάρξει δυνατότητα να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 2 του κανονισμού μας. Και πάλι, ε, δεν είναι αυτή η τελική ψηφοφορία. Δεν ψηφίζουμε την έκθεση. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική ψηφοφορία όμως για τροπολογίες βάσει του άρθρου 70 παράγραφος 2 του κανονισμού μας. Επίσης, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι κάποια μέρη αυτών των εκθέσεων, για να τις χαρακτηρίσω έτσι, ξέρετε τι εννοώ, θα ψηφιστούν μετά το καλοκαίρι, ας πούμε, αιτιολογικές σκέψεις, δεν θα ψηφιστούν σήμερα. Ε, και κάποια άλλα στοιχεία των τροπολογιών που δεν μπορούν να ψηφιστούν για διάφορους λόγους. Άλλες ε, είναι τεχνικές τροπολογίες που δεν έχουν οριμάσει ακόμα. Άλλες ε, συνδέονται άμεσα με το ε, θέμα της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού κανονισμού που ακόμα εκρεμεί και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια μετά τις ερηνές διακοπές. Λοιπόν, για διάφορους λόγους δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τα πάντα σήμερα. Παρόλα αυτά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ψηφίσουμε όσο γίνεται περισσότερα και επίσης τα άρθρα κυρίως που δίδουν τη βάση για τη διαπραγματευτική εντολή. Δεν είναι οι τελικές προτάσεις, οι τελικές ε, οι οριστικές αν θέλετε, αλλά δίνουν την εντολή. Λοιπόν, Αφού ψηφίσουμε το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα σας προτείνω να εγκρίνουμε τη διαπραγματευτική εντολή και θέλω και την υποστήριξή σας και να σας ενημερώσω ότι θα υπάρξει ξεχωριστή διαπραγματευτική ομάδα για κάθε τμήμα του κανονισμού. Επίσης να σας ενημερώσω ότι η διάσκεψη του Προέδρου του Κοινοβουλίου μας αποφάσισε την 5η Ιουλίου συγκεκριμένα οι εργασίες του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ και οι αντίστοιχες νομοθετικές ε, προτάσεις και το πλαίσιο θα πρέπει να συντονιστούν. Και μας ζητήθηκε ε, από τις επιτροπές να διαπραγματευτούμε, αλλά να μην ε, ολοκληρώσουμε τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, ούτε να κάνουμε deal, διάφορες συμφωνίες για μεμονωμένους τομείς πολιτικής και να σεβαστούμε την αρχή ότι τίποτα δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα. Υπάρχει και η δική ομάδα στην οποία προεδρεύει ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε. Θα ήθελα επίσης να σας θυμίσω και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό αν θέλετε στις συζητήσεις σας ότι ε, τους τελευταίους εννέα μήνες από τότε που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έστειλε τις νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο, είχαμε δέκα συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Επανειλημμένα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις νομοθετικές προτάσεις και επίσης 11 ομάδες εργασίας ασχολήθηκαν στις συνεδριάσεις τους, 11 συνεδριάσεις δηλαδή, με αυτό το θέμα. Και ε, αμέτρητες ήταν οι συνεδριάσεις των σχεδόν εισηγητών, των πολιτικών ομάδων, το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι τεράστιο το έργο που κρύβεται από πίσω. Όχι μόνο η γραμματεία και εσείς, ε, οι βοηθοί σας, οι πολιτικές σας ομάδες έχετε ξαγρυπνήσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας μέχρι να μπορέσουμε να ψηφίσουμε το σχέδιο εκθέσεων όπως έχουν κατατεθεί από τους ε, ε, εισηγητές το τέλος αυτής της διαδικασίας. Με όλα αυτά τα εισαγωγικά που σας είπα λοιπόν θα ήθελα να πω ότι τα άρθρα που συνδέονται με τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν θα τα ψηφίσουμε αλλά το έχει φροντίσει η γραμματεία Yes, I understand, but you have taken care of, this, so you... Ναι, ναι, μα το φροντίσατε έτσι και θα μας το επισημαίνετε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Μην τυχόν και ψηφίσουμε πράγματα που δεν κάνει τώρα πια, ε, τόσο νωρίς. Ε, και ένα τελευταίο που θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε πριν πέρασουμε στην πρώτη ψηφοφορία είναι ότι έλαβα ένα αίτημα για να το χαρακτηρίσω έτσι, η πρόταση, η υπόδειξη ότι μπορούμε αν μπλοκ να ψηφίσουμε κάποιου συμβιβασμού διότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Αλλά γι' αυτό θα χρειαστώ την συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων. Ορίστε κυρία Σρότερ, έχετε σχέση εσεί με αυτή την πρόταση, θα μπορούσατε να μα πείτε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Να μιλήσω γερμανικά. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία. Ε, είναι πολύ καλά καταρτισμένος ο κατάλογος ψηφοφοριών. Ε, τον πήραμε χτες το βράδυ. Ήταν πολύ καλή, πολύ σκληρή δουλειά. Άντεξαν και έκαναν πραγματικά σπουδαία δουλειά. Ευχαριστώ τη Γραμματεία. Αλλιώς θα πρέπει να επικρίνω τη διαδικασία, διότι... δεν έλαβε χώρα η διαπραγμάτευση ε, όπως έγινε σε άλλες επιτροπές που γνωρίζω ότι έγινε και που υπήρχαν δυνατότητες να γίνει και εδώ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Μια μικρή πολιτική ομάδα έκανε μεγάλη προσπάθεια να δουλέψει ε, επί της ουσίας στη διαδικασία αυτή, να βάλει το λιθαράκι της. Τελικά είναι αδύνατο να δούμε τι προέκυψε και αν θα συμφωνήσουμε. Έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορία ε, τελικό που τον πήραμε τα μεσάνυχτα. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε πια. Και ε, το είπαμε και στις διαπραγματεύσεις. Δεν επιτρέπεται γιατί και επί της ουσίας θέλουμε να εργαζόμαστε κανονικά και να ξέρουμε τι ψηφίζουμε και να μην ψηφίζουμε μόνο κάποια νούμερα ε, τυφλά. Είμαστε κατά αυτής της πρόταση λοιπόν των ε, unblock ψηφοφοριών και δεν ε, το έχει τώρα σημασία ε, τόσες ψηφοφορίες που έχουμε, να κάνουμε και 10 παραπάνω δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά ξέρουμε όμως την ουσία τι ψηφίζουμε και τι βγαίνει. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Τώρα η μόνη απόφαση που σας ζητώ να με βοηθήσετε να πάρουμε και να πάρω εξ ονόματός σας είναι εάν θα ψηφίσουμε του συμβιβασμού. on Όχι, η πράσινη είναι κατά. Ναι, ναι, το καταλάβαμε αυτό. Ε, ο κύριο Πανίστερα. Δεν θα αρχίσει η συζήτηση όμως. Όχι, όχι, όχι. όχι. Έχουμε αρκετά θέματα να ασχοληθούμε. Ε, ένα σχόλιο μόνο. Το κείμενο που διανεμήθηκε την περασμένη εβδομάδα, που εστάλει, μια στιγμή ένα σχόλιο. Έλεγα, στείλαμε ένα κείμενο την περασμένη εβδομάδα για τους συμβιβασμούς και είχε συζητηθεί από τις πολιτικές ομάδες με τους σκιώδεις και χτες είχαμε τελευταίο έλεγχο και χτένισμα. Έχω σχόλια σε δύο σημεία που διαφέρει το κείμενο από εκείνο που είχε αποσταλεί και θα σας το ανακοινώσω ποια είναι τα μικρά που έχουν αλλάξει διατυπώσεις. Είναι πάρα πολύ τεχνικά αυτά. Κατά τα λοιπά το κείμενο παραμένει ως έχει και χτες και προχτές και τις προηγούμενες μέρες που το είχατε. Και το συζητήσαμε. Δεν υπάρχουν εκπλήξεις τίποτα μέσα σε αυτό το πακέτο. Αυτό ήταν το αρχικό μου σχόλιο. Κύριε Σιμάζε. Κοιτάξτε, είπαμε συζήτηση δεν θα κάνουμε. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής ε, και το προσωπικό των πολιτικών ομάδων και τους βοηθούς μας γιατί έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να σας πω ότι εκπλήσωμαι από το αίτημα. Τελευταία στιγμή δεν μπορείτε να μας ζητάτε να ψηφίσουμε μαζί κάποιους συμβιβασμούς ε, αμπλόκ αφού έχουμε ε, κάνει καταλόγους ψηφοφορίας από κοινού. Αυτό συμφωνήθηκε. Λοιπόν, να τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Διαφωνεί και η δική μας ομάδα. Πόσο μάλλον που είναι ξέφρενοι οι ρυθμοί τώρα στην ψηφοφορία. Εντάξει, ωραία. Ε, οι πράσινοι το πρότειναν και ήταν σαφές ότι η κυρία Σρότερ απέσυρε την πρόταση αυτή, οπότε δεν χρειάζεται πια να τη συζητήσουμε. Ε, τι έκανα? Δεν, ζήτησα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ, λέει η κυρία Σρότερ. Εντάξει, να το συζητήσουμε μετά αυτό. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Συγγνώμη. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα κάνουμε block vote. Χτες στις διαπραγματεύσεις αρνηθήκαμε. Και σήμερα αρνηθήκαμε. Δεν ζητήσαμε ποτέ να κάνουμε block ψηφοφορίες. Η, κυρία Κρέλ γι' αυτό. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ, ψυχραιμία. Εάν μια πολιτική ομάδα, οι δύο είναι κατά, Εντάξει, εχθές με τους σκιώδει συζητητές έγινε μια πρόταση που δεν ήρθε από τους πρασίνους και προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και να την ελαφρύνουμε. Εάν δεν συμφωνούν οι ομάδες, Καλώ δεν υπάρχει πρόβλημα. Ψηφίζουμε όπως το προβλέπει ο κατάλογος ψηφορία. Κανένα πρόβλημα. Thank you. So decided. So there's no... Εντάξει, ούτως αποφασίζεται, έληξε αυτό το θέμα. Κύριε Τσέλερ, γι' αυτό θέλετε. Με ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένης της κατάστασης, δεν μπορώ και εγώ να σας βοηθήσω για να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Ωραία, θα ψηφίσουμε, όχι αμπλόκ. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να ζητήσω στο συμβιβασμό 50, στη συμβιβαστική τροπολογία, να ψηφίσουμε το κάθε τμήμα ξεχωριστά για την 50 συμβιβαστική. Όταν φτάσουμε εκεί, θα σας πω ποιες θα είναι κατά τμήματα, ψηφοφορίες, χωριστές. Ε, για να τα πω τώρα, για να μην μιλήσω στη συνέχεια. Ε, η γραμματεία έστειλε ένα πολύ σαφές μήνυμα στις 5 Ιουλίου και έδινε την ε, προθεσμία ε, για τα αιτήματα για χωριστέ ή κατά που ήταν τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα. Οποιοδήποτε αίτημα κατατέθηκε εκ πρόθεσμα δεν μπορεί να ε, γίνει δεκτό και δεν θα δώσουμε συνέχεια. Επιπλέον, αυτά που ακούμε σήμερα να ζητάτε είναι εκ και δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Πάμε. Τροπολογία παριθμών 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 357 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 358 Στο μεταξύ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι επειδή είναι πάρα πολύ περίπλοκη αυτή η ψηφοφορία, από καιρού καιρό θα χρειάζεται η γραμματεία να κάνει κάποιες επαληθεύσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στη σελίδα 4 και ψηφίζουμε την 23 της Επιτροπής Απασχόλησης. Έμπλη 23. Υπέρ. Στη σελίδα 4 κάτω. υπέρ. Περιμένω μια στιγμή γιατί ψάχνονται οι συνάδελφοι. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 24 της Επιτροπής Απασχόλησης στη σελίδα 6. Έμπλο 24. Ψηφίπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25 στην ίδια σελίδα ε, της Επιτροπής Απασχόλησης κάτω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σαφώς. NV11 στην επόμενη σελίδα. Η 11 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ερχόμαστε στη συμβαστική υπαριθμών 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στη σελίδα 10 παρακαλώ. Τροπολογία 387 που είναι ταυτόσιμη με την 28 της Επιτροπή Απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Στη σελίδα 11 η 17 της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Κοντ 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ή 20. Σε ποια σελίδα είναι η 11, κάτω-κάτω. Η 20 της Επιτροπής Βιομηχανίας. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 393 στη σελίδα 11, λίγο πιο πάνω. Θεωρείται ότι έχει ψηφιστεί πριν την Ήτρα και, και την κοντ. 393 με τη σειρά αυτή. Η ψήφη υπέρ. Στη σελίδα 11. Η ψήφη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Άρα η 17 της ε, ε, Επιτροπής Ελέγχου καταπίπτει και η 20 της Ήτρα καταπίπτει. Διορθώνουμε λοιπόν τη ψηφοφορία που κάναμε προηγουμένως. 394 στη σελίδα 12. Υπέρ τη 394. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. Η 30 της Επιτροπής Απασχόλησης στην ίδια σελίδα υπέρ. Κατά. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν καταλαβαίνω τίποτα, γιατί τα ε, νούμερα δεν συμπίπτουν. Δεν καταλαβαίνω πού βρισκόμαστε. Μα δεν μπορούμε να ψηφίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. γιατί υπάρχουν τροπολογίες που πρέπει να ψηφιστούν σύμφωνα με τις συζητήσεις που έγιναν με τους Κεώδης και τη Γραμματεία που μπορεί και πρέπει να ψηφιστούν ως προσθέσεις στις συμβιβαστικές και υπάρχουν τροπολογίες που που καταπίπτουν όταν υιοθετηθεί ένας συμβιβασμό. Γι' αυτό πάμε σιγά σιγά. Ναι, αλλά εγώ είμαι συνηθισμένος να ψηφίζω και θέλω να καταλαβαίνω τι ψηφίζω. Διαφορετικά δεν ψηφίζω. Πρέπει να καταλαβαίνω τι γίνεται, τι ψηφίζουμε, γιατί διαφορετικά δεν θα ψηφίζουμε. Wait a minute, Mr. De Angelis, can, can we... Μισό λεπτό κύριε De να μπορούμε να εξηγήσουμε στους συναδέλφους κύριε Ολενίτσα και μετά η κυρία Κρέλα. Ίσως εγώ μπορώ να βοηθήσω. Έχουμε έναν κατάλογο που είναι ελαφρώς διαφορετικός από αυτό που έχετε εσείς. Βασικά σημαίνει ότι όταν ε, μιλάτε για μια συγκεκριμένη σελίδα, εμείς είμαστε αλλού για αλλού και βλέπουμε διαφορετικές τροπολογίες. Μήπως λοιπόν καλύτερα να μην καν για ποια σελίδα μιλάτε και να μιλάτε μόνο για το νούμερο της τροπολογίας. Θα είναι πιο εύκολο έτσι. Yes, ε, ε, Ναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι από ό,τι φαίνεται η δική μου ομάδα έχει τυπώσει διαφορετικά τον κατάλογο ψηφοφορίας από αυτό που έχετε εσείς ή και εγώ. Και ε, επειδή ε, έχουμε πρόβλημα με την αρρύθμιση των σελίδων, αν θέλετε να πείτε το άρθρο. Αλλιώς να κοιτάει η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, τη σειρά των τροπολογιών χωρίς να κοιτάει σελίδες. Ναι, δεν έχω πρόβλημα να, να πάω πιο, πιο σιγά αλλά δεν μπορούμε να αποφεύγουμε γιατί υπάρχουν ε, τροπολογίες ε, που είναι συμπληρωματικέ και άλλες που καταπίπτουν. Πρέπει δηλαδή να συνδέονται οι τροπολογίε με τις συμβιβαστικές και γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο. Αλλά ναι, θα τα πω λίγο πιο αργά. Θα τα πούμε πιο αργά και δεν θα μιλάμε για σελίδες, θα μιλάμε για, για Λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε. So we move now to Περνάμε λοιπόν στην 395. που είναι μετά από την 30 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3 τώρα. Μετά από την τροπολογία 395 σε όλους τους καταλόγους. Ποιοι είναι υπέρ της συμβιβαστικής 3, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. So now we move to employment 33. Which is inside compromise 3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 θα πάρει πιο πολύ ώρα από ό,τι συνήθω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αλλά έχουμε πάνω από 2.000 τροπολογίε. Βρήκατε λοιπόν την τροπολογία τη Επιτροπή Απασχόληση υπαριθμών 33. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά έχουμε την 421. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια εικοσιεπτά υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 439, δύο-τρει σελίδε πιο κάτω. 439, ουτζία. υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 442 που ακολουθεί. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 443 ναι, έχει καταπέσει. Ναι, ναι. Ναι. Έχουμε τώρα την τροπολογία 37 της Επιτροπής Απασχόλησης που είναι προσθήκη. 37 απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 444 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 41 της Επιτροπής Απασχόλησης απορρίπτεται και πάμε στην συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τετρακόσια 466 ε, με συγχωρείτε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ήτρε 27. Ήτρε 27. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 10 που είναι παρακάτω. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. There Φτάνουμε στην, 44 της Επιτροπής Απασχόλησης. Και είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 47. της Επιτροπής Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. one, two, three pages, everything pages. So I think So we move to compromise. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε ένα σωρό σελίδες και μάλλον όχι ένα σωρό, φτάνουμε γρήγορα στη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβιβαστική 9. Ποιοι είναι υπέρ της 9. Οι υπόλοιπες έχουν καταπέσει. Κατά αποχές εγκρίνεται. Mm. So we now, after four or five pages uh, of... Μετά από 4-5 σελίδες ακόμα διάφορες τροπολογίες που έχουν καταπέσει, φτάνουμε στην τροπολογία 550. 550. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κάτω από αυτήν έχουμε τη συμβαστική 10. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έχουμε πάλι αρκετές σελίδες. We go to 562. Πάμε στην 562. 562. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 με την 11 της ΠΕΣ και την 583. Μπορούμε να ψηφίσουμε. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Okay. One, two, three pages of falling amendments and 592. Περνάμε στη 592 και ψηφίζουμε για αυτήν. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Then again we have falling amendment. Και πάλι έχουμε σελίδες με διάφορες τροπολογίες που καταπίπτουν. Και φτάνουμε στην 622. Did you find it? Who is in favor? Τη βρήκατε, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται ήταν συμβατή και με την 60 της Επιτροπής Απασχόλησης. Yeah. Colleagues have to check. No, we we have to be patient because we have to... Υπομονή παρακαλώ για να τα κάνουμε σωστά. Okay, so employment 60 is not όχι. Η 60 δεν είναι ταυτόσιμη, είναι απλώς συμβατή. Πρέπει να ψηφίσουμε και την 60, λοιπόν, της Επιτροπής Απασχόλησης, που είναι κάτω από την 622. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. So we move now to 627. 627. Προσθήκη. Ποιοι είναι υπέρ. 6.27. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. So we move to compromise 12. Περνάμε στην συμβιβαστική 12. Τι λέτε 631, 631 καταπίπτει. Πάμε στη συμβαστική 12. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έξι Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έκον 12. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. And we go to compromise 14. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Five, at least six pages of calling amendments. seven. So we move to 691.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 Ψηφίζουμε την 691. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι ίδια με την 693. It's not adopted, it's withdrawn. So we vote employment 74. Απασχόληση 74. Απασχόληση 74. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60. Who is... 60. Υπέρ,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 We one, Μισό λεπτό γιατί επιδείξαμε μια τροπολογία. Πρέπει να ψηφίσουμε για την 677. Πάμε στην 677 λοιπόν. Τι βρήκατε. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Ωραία. Ήτρε 56. Ήτρε 56. Υπέρ, κατά, αποχές. απορρίπτεται. Απασχόληση 75 έχει καταπέσει. 705. Ψηφίζουμε την 705. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 706 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 77 της ε, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Καταπίπτει. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά εποχές δεκτή. Ερώτηση είναι κυρία Ματσόνη. Έχω μια αμφιβολία όσον αφορά την πρόταση στη συμβαστική, γιατί ένα τμήμα είναι πιο έντονα αρμένο. Θέλω να καταλάβω αν αυτό το κομμάτι που σχετίζεται με την παράγραφο 4 δεν υπάρχει πια στη συμβαστική πριν να ψηφίσουμε. Ναι. Λοιπόν. Υπήρχε ένα κείμενο που δεν κόλλαγε εκεί και που ήταν μάλιστα από το αρχικό κομμάτι αλλά τώρα πλέον δεν είναι μέσα αυτό στο σημείο 4 έχει φύγει το κείμενο Without paragraph... Χωρίς, χωρίς την, την παράγραφο 4. Ναι, καλά τα λέω. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα το ξεκαθαρίσαμε. Ε, ούτως ή άλλως θετικά ψηφίσαμε. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Περνάμε στην ε, Επιτροπή Απασχόλησης που είναι αρκετές σελίδες παρακάτω. 80 από την Επιτροπή υπέρ καθά, αποχές απορρίπτεται rejected it was rejected 62 amendments 62 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Which one? So we move to 736. 736. Υπέρ. 114 σελίδα. Κατά αποχές απορρίπτεται. 737 υπέρ. κατά αποχές απορρίπτεται η επόμενη καταπίπτη ...739 προφορική τροπολογία. Είναι κάποιος κατά? Παρακαλώ, κύριε Πίπερ. Θέλω να αποσύρω αυτή την τροπολογία, λέει ο κύριος Πίπερ. Μάλιστα. Δεν την ψηφίζουμε λοιπόν. «739 αποσύρεται». Περνάμε σε δύο σελίδες παρακάτω. 21 της Επιτροπής Ανοιχτού του Προπολογισμού. 116, 116 σελίδα. 21 της Επιτροπής Ένωσης ταυτόσιμη με την 59 της Ήτρε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 της ΕΚΟΝ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 17. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. 767. Δύο-τρεις σελίδες παρακάτω. 765. Με συγχωρείτε. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 771 δύο σελίδες παρακάτω υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται τραν 22 υπέρ ακριβώς από κάτω καταπίπτει Α, μάλιστα είχε υιοθετηθεί η προηγούμενη οπότε καταπίπτει είναι καλά λέτε 776 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 τώρα τι θέλετε έγινε δεκτή η συμβαστική μα δεν, ναι, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εφτά, οχτώ, εννιά. Μαζί με την 92 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 791 από κάτω υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 799 υπέρ κατά αποχές δεν ξέρω νομίζω ότι απορρίφθηκε να επαληθεύσουμε 799 Είναι κάποιο παραπάνω από το ΕΛΚ, παρακαλώ να βγάλει την τη κάρτα. Εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Μάλιστα. Δεν ξέρω. 37 ε, κατά. 93 της απασχόλησης ε, Συν 132 του ΕΛΚ 93 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να την απαληθεύσουμε δεν ξέρω κάπου εκεί στα ορεινά κάποιος θέλει να επαληθεύσει αλλά δεν, δεν ξέρω αν βουλευτές εκεί πίσω 800 808 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 825 εικοσιπέντε συνάδελφοι 137 σελίδα Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 825. Ναι, μάλιστα δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι. Απορρίφθηκε. Για τον Λαμπέρ το κάνουμε. 829 829 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή έχουμε τα χρηματοοικονομικά μέσα, δεν τα ψηφίζουμε όπως συμφωνήσαμε. που είναι πολλές σελίδες και περνάμε στην 933 που είναι τη βρήκατε 933 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Καταπίπτει, καταπίπτει. 104 της Επιτροπής Απασχόλησης. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή. και περνάμε στην επόμενη συμβιβαστική με παρθμόν 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή Πρέπει, πρέπει να αντεπαληθεύσουμε, συνάδελφοι, για να είμαστε σίγουροι. Εκατόν δώδεκα της Επιτροπής Απασχόλησης. Σελίδα 161. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Καμιά φορά οι προτάσεις σας δεν είναι σωστές, πρέπει Ό,τι ακούγεται από να το ελέγχουμε. 9.76 περνάμε τώρα ακριβώς μπροστά από την επόμενη συμβαστική 9.76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 35 105 ναι ναι υπέρ κατά αποχές δεκτή μπορώ να πάω στη συμβαστική 35 επιτέλους ναι υπέρ κατά αποχές δεκτή ακολουθούμε και τη γραμματική σας. Λοιπόν, συμβαστική 36 υπέρ κατά εποχές δεκτή. 1000 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. Πενήντα της γυναικών. 50 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 38 υπέρ Συμβαστική 38 κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 40 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «126 Επιτροπής Απασχόλησης» ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 41 υπέρ 41 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 της Επιτροπής Απασχόλησης. 132 Στο μεγάλο κατάλογο είναι στη σελίδα 178, στο τόμο αυτό. 132. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1054. 1054. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1055. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβιβαστική 42 είπε Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 1058. Από κάτω. Υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1063 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 1064 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οικονομική 21. Σελίδα 182 Λάμπερτ. Ε, υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 135 της απασχόλησης. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 1075 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1076 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται από ό,τι βλέπω 1077 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 46 τώρα λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 το λέω για τον Βανίστε Ρόι. 30 ε, ε, ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού. Χίλια εκατόν Χίλια Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1119 λίγο πιο κάτω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 52 της Επιτροπής Γυναικών υπέρ αμέσως μετά είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεν θα ψηφίσουμε γιατί είναι του δημοσιονομικού κανονισμού οι επόμενες και προχωρούμε. Και η 1128 το ίδιο, οπότε θα την ψηφίσουμε και η 40 της ΕΜΒΗ μπορεί να ψηφιστεί. Την έμβη 40 τι θα την κάνουμε. Θα την ψηφίσουμε. ΕΝΒΗ 40. 40 της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Για το ΕΛΚ είναι σελίδα 190 στο χωτρό κατάλογο. Μπορώ να σας λέω τις σελίδες, αλλά η Κωνσταντζε θα μπερδευτεί. 190 λοιπόν, σελίδα υπέρ κατά αποχές, απορρίφθη. 11.30 ε, υπέρ κατά, αμέσως ε, μετά είναι, στην αποχές εγκρίνεται 1135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα μια στιγμή Μια στιγμή κάνει κάτι επαληθεύσει η γραμματεία και χρειάζεται προσοχή εδώ. Τι λέτε, μπορούμε να ψηφίσουμε την 123. Μάλιστα, είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται η 30 του προϋπολογισμού. Α, είναι πακέτο, όλα αυτά είναι ταυτόσημα, δεν χρειάζεται. «1141» στην επόμενη σελίδα. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, 1143 ε, υπέρ. 1143. Όχι. Α, όχι, ναι, και πάλι το δημοσιονομικό κανονισμό δεν μπορεί να ψηφιστεί. Να μου το λέτε, σας παρακαλώ. Τελικά ψηφίζουμε 11.43. Δεν ξέρω, δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Μια στιγμή να το κοιτάξουν οι συνάδελφοι. 1148, 1148, στη σελίδα 193, στο μεγάλο κατάλογο. Υπέρ της 1148 κατά αποχές εγκρίνεται. «1150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». 1154. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι ταυτόσιμη με μερικές άλλες. Μια στιγμή για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. 31 της Επιτροπής Ελέγχου προπολογισμού. Εκεί είμαστε. Όχι. Στην 32, όπου, όπου και αν βρίσκεται αυτή. Είναι πιο κάτω. Η 31, όχι. Α, όχι, στην 31 της Επίτροπης Ελέγχου είμαστε. Υπέρ κατά αποχές ναι, απορρίπτεται. Τώρα πάμε στην 32 της Επιτροπής Ελέγχου. Κοντ 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1173 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η επόμενη καταπίπτει 1176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εκείνη συμβατή με την 33 της Επιτροπής Ελέγχου. Και τώρα... 77. ψηφίζουμε. έχετε δίκιο. Ε, υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν η, 33 αυτή της Επιτροπής ε, Ελέγχου. Ναι, πρέπει να επιβραδύνουμε λίγο, ζητώ συγγνώμη. 1177, we can vote 1177. 1177 υπέρ κατά αποχές όχι. Απορρίπτεται. Είστε σοβαροί. Α, τώρα έχετε διάθεση ήδη για αστεία. Πολύ νωρί σα ήρθε. Λοιπόν, έλεγχος. Γιατί 34, όχι ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές, απορρίπτεται η 34 της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού. Ήτρε 76. Είναι μέσω μετά Λαμπερτ. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. ΠΕΣ 20 της Επιτροπής Αλίας υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1186 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1189 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται NV41 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται απασχόληση 144 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται NV42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 145 απασχόληση καταπίπτει αν εγκριθεί 144, δυστυχώς 144 περίφθη, άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 145 της Επιτροπής Απασχόλησης. Υπέρ. Όχι. Καλά. Ας μην την ψηφίσουμε, εσείς ξέρετε. Άρα, πάμε, δεν θα την ψηφίσουμε τότε. Καταπίπτει, εν πάση περιπτώσει. Ωραία. Και 146, ε, πάντα της Επιτροπής Απασχόλησης, οπότε ερχόμαστε στη Γεωργία. Όχι, όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό. Πάμε στην 1199. Ως προσθήκη. Στη 201, ε, σελίδα 201. 1199 ως προσθήκη στο συμβιβασμό 48. 1199. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σελίδα 203, 1203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική τώρα νομίζω όχι όχι ακόμα πριν τη συμβιβαστική έχουμε κάτι άλλο τη 1208 1208 την ψηφίσαμε. Υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Συμβαστική 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 50 υπέρ. Ναι, κύριε Τσέλερ. Ναι, ναι, εντάξει, περιμένουμε, εντάξει. Would like to say something probably auf Deutsch. Ο κύριος Τσέλερ θα πει κάτι μάλλον στα γερμανικά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε ζητώ σε αυτή τη συμβαστική τροπολογία ε, χωριστή ψηφοφορία ε, στην παράγραφο 1 στο β λατινικό και ε, το σύνολο της παραγράφου 3. Κατά τμήματα λοιπόν ψηφοφορία, όχι ολόκληρη της συμβαστική. Ναι, για το τυπικό του θέματος όμως, όπως σας είπα στην αρχή, εξέπνευσε η προθεσμία. Έπρεπε να το είχατε ζητήσει εμπρόθεσμα αυτό το πράγμα. Τώρα δεν μπορώ να δεχτώ τέτοιο αίτημα για ψηφοφορία κατά τμήματα. Λυπάμαι, γιατί απορρίψαμε πάρα πολλά αιτήματα που κατατέθησαν πρόθεσμα και δεν μπορώ να δεχτώ το δικό σας. Κύριος Πίπερ. Ποιος από τους συναδέλφους εδώ γνώριζε αυτή την προθεσμία. Τουλάχιστον τα συνήθη μέλη τα απλά μέλη της Επιτροπής δεν είχαν αυτή την πληροφόρηση. Δεν θα ήταν δίκαιο και σωστό τώρα να δεχθούμε αυτή την ε, υπόθεση που ζητάει ο κύριος ε, γιατί είναι και οι ενδιάμεσες κατηγορίες και οι ποσοστώσεις που δεσμεύονται από το κοινωνικό ταμείο ε, και άλλα τέτοια και με τις βατικές περιφέρειες μας αναγκάζουν ε, συνολικά να δεχθούμε ή να απορρίψουμε αυτή την τροπολογία. Κυρία Χιούμπνερ, στο δικό σας χέρι είναι. Εσείς μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα ψηφιστεί ή όχι. Όχι η Επιτροπή, εσείς το αποφασίζετε αυτό. Ευχαριστώ, η Κωνσταντζε. Κρέ. Ναι, θα παρακαλούσα θερμότατα, όπως είπε και ο Μάρκος Πίπε, να δούμε αυτό το συμβιβασμό. Ε, είναι πάρα πολύ ε, μεγάλο. Είναι μια συνολική ε, υπόθεση αυτή και θα πρέπει να ψηφιστεί συνολικά γιατί είναι συνολική και η διαπραγματευτική εντολή. Στα επιμέρους θα επανέλθουμε στην Επιτροπή και θα ξανασυζητήσουμε μετά τον τριμερή διάλογο με το Συμβούλιο. Αλλά σας παρακαλώ να το δούμε ως ένα πακέτο, ως μία δέσμη συμβαστική. Γιατί αν αρχίσουμε να ξυλώνουμε τώρα την πρόταση και επιτρέπουμε ψηφοφορίες χωριστές, τότε θα βγει ο καθένας και θα πει και εγώ θέλω το δικό μου θέμα να ψηφιστεί χωριστά. Όχι. Νομίζω ότι είναι πραγματικά ισορροπημένη αυτή η συμβαστική πρόταση και την προτείνουν και οι δύο συνεισηγητές. Ναι, ο κύριος Γκοντμάνης. Μια στιγμή να θυμίσω, επειδή αμφισβήτησε την πληροφόρηση ο κύριος Πίπερ και ο Μάρκος ε, και ο Γιώχημ ε, Τσέλερ είναι στο κατάλογο παραλήπτων ε, στο μήνυμα το ηλεκτρονικό που έστειλε η γραμματεία για την προθεσμία ότι έλεγε στις 6 ώρα το απόγευμα της Δευτέρας 9 Ιουλίου και μάλιστα το mail αυτό εστάλει στις 5 του μηνός Ιουλίου. Σας ενημερώνω για τα τυπικά πώς έγινε η πληροφόρηση αυτή και γιατί δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Είναι κάτι έκτακτο, εκπρόθεσμο και δεν είναι παραδεκτό. Παρακαλώ δεχτείτε τον κανόνα που υποχρεώθηκαν να δεχθούν και άλλοι συνάδελφοι. Ποιος ήθελε ο κύριος Γκοντμάνης, παρακαλώ. Θα ήθελα κι εγώ να υποστηρίξω ε, το να μην γίνει χωριστή ψηφοφορία. Ήταν τεράστιο το πρόβλημα να φτιαχτεί αυτός ο συμβιβασμός, σε πάση περιπτώσει. Και γιατί χρειάζεται αυτή η συμβαστική πρόταση, γιατί... Ε, από οικονομικής πλευράς θα είναι το βασικό μας ατού απέναντι στο Συμβούλιο. Αν χωριστούμε εδώ, θα ήταν μεγάλο το πρόβλημα να συζητήσουμε. Ε, είναι τα πάντα, ιδιαίτερα απομακρυσμένε, διαφορετικέ περιφέρειε, ασφαλιστικά ε, ε, δίκτυα ασφαλεία. Αν αρχίσουμε να το ξυλώνουμε αυτό, δεν θα πετύχουμε τίποτα. Και σε καμία περίπτωση. Και εγώ θα παρακαλούσα να μην διχαστούμε από αυτού. Ευχαριστώ. Άλλο σχόλιο. Δεν βλέπω υποστήριξη ο κύριος Τσέλερ. Τότε ζητώ να ψηφίσουμε με το μηχάνημα ονομαστικά. Ναι, μάλλον. Φαντάστηκα ότι κάποιος σας ζητούσε έλεγχο. Ο Λάμπερτ Βανίστερ Ρόι. Συγγνώμη, πρέπει... Ε, σας είπα ότι θα ξανάρθω όταν έχω διευκρινίσει μια λεπτομέρεια. Είναι στο συμβιβασμό 7 η διατύπωση να βγει είναι κάτι που λέει ενδεικτικά. Πώς το προφέρουν αυτό. Indicatively. Ενδεικτικά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, άλλο, για άλλο συμβιβασμό μιλάς εσύ. Ναι. Και για... Στο 50 δεν είναι. Στο 50 είναι. Είναι στο 50, ε, στο 7 όμως. να βγει αυτό το, η αναφορά στο ενδεικτικό. Περίμενε, πού είναι αυτό όμως. Είναι πρόταση για προφορική τροπολογία αυτό, διαφωνεί κανείς. Η κυρία όχι δεν θέλουμε άλλες προφορικές τροπολογίες. Ορίστε, διαφωνούν οι πράσινοι, δεν υπάρχει αυτή η τροπολογία και προχωρούμε. Ηλεκτρονικά, έτσι από την αρχή για να μην έχουμε προβλήματα. Ψηφίζουμε το συμβιβασμό 50 ηλεκτρονικά όπως ζητήθηκε. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. We are voting for the compromise. Το συμβιβασμό ψηφίζουμε, όχι για συζήτηση. Το συμβιβασμό, έτσι, τη συμβαστική τροπολογία 50. Τρεις ακόμα δεν έχουν ψηφίσει και περισσεύει ένας από το ΕΛΚ. Εντάξει, πέρας. Ψηφίσατε όλοι. 41 υπέρ, 5 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν ο συμβασμό υπαριθμό 50. Και προχωρούμε. 12. 12.46 είναι αυτό που πάμε τώρα. Σελίδα 216 στο μεγάλο κατάλογο. Ναι, το βρήκα, λέει ο κύριος Φανίσερε. Μπράβο σου, εγώ ακόμα δεν το βρω. 1246 ε, υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε την ITRE 32. Ε, Ελέγχουμε τις τροπολογίες που μπορεί να την έχουν κάνει να καταπέσει. Maybe somebody is faster with finding how we voted on 1301, then that would help the colleague. Αν κανείς θυμάται τι κάναμε στην 1301 Όχι, θα σας αφήσω να πάτε για φαΐ. Μην χωριέστε. Αλλά δεν θα σας καλέσω. So we can vote.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 Um, Τα καλά νέα είναι ότι τόσο πολλά καταπίπτουν όταν ψηφίσουμε μια ε, συμβιβαστική. Απασχόληση 153. Απασχόληση 153. Περ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 44-49 πέρα αποχε... Ε, κατά αποχές απορρίπτεται 13-34 13-33 συγγνώμη διορθώνω η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1336 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Unfortunately, not to the end of the Yeah, 1351. 1351 in favor. 1351. Μισό λεπτό γιατί η Νταϊάννα δεν είναι ευχαριστημένη.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 Τροπολογία 1, 3, 4. Αλλά μπορούν ηλεκτρονικά να το κάνουν πολύ γρήγορα. No, we have to be sure, yeah. But... Όχι, πρέπει να είμαστε βέβαιοι. They, they know what they are doing. They... Uh, okay, so it's just uh, under the compromise 52. Συμβιβαστική 52.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 1351, I think we, we have to vote what 13 we have to vote now 1351. 1351. 1351. Ποια είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Now we vote employment one. Ψηφίζουμε την απασχόληση 159 στη σελίδα 246. 159. In favor. 159 Επιτροπής απασχόληση υπέρ κατά ε, αποχέ απορρίπτεται. Μα έχουμε συμφωνήσει τώρα σε αυτό. Δεν ξέρω γιατί έχετε διαφορετικές σελίδε. Θα έπρεπε να έχετε τις ίδιες σελίδε με τον Πρόεδρο. not asking anyone. 1384. 1384. 1384, δεν θα λέω τη σελίδα. 1384 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεκατρία 1392 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Χίλια τετρακόσια 1408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 96 είναι η επόμενη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν επτά. Ε, συγγνώμη, 14-17. Υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. Απασχόληση 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14-18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά δεν ψήφισαν όλοι 141 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14.32 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14.33 Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 14.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1436 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κοντ 50 υπέρ... Όχι, καταπίπτει γιατί εγκρίθηκε η 1434. Συμβιβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1441 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1447 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 100. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 101. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβεβαστική 54. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 55, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε στην 1470. 1470, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σεμβαστική 56 υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται. Απασχόληση 178. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. FAM 58. FAM 58. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήτρε 102, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 1488, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 1489 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1491 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβαστική 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται We go on. Just go on. To 1520, no? Yes. 1520. 15-20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15444. 1544. 1544 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1546 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1548 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1551 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1553 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1554 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1557 υπέρ αποχές εγκρίνεται 1558 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 60 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται And then we move to 1578. It's page 286. 1578. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 193. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται γυναίκες 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γυναίκες 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Απασχόληση 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1590 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. False. 1628, 1628. Sorry, 1628. Yes, 1628. it's page 295. 1628. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φάμα 62 υπέρ κατά αποχές απο, ε, απορρίπτεται. 16-29 16-29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16.30. Είναι κανείς κατά. Όχι. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16.31. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Επασχόληση 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 16.32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ήτρε 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 163% υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 16-19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 16.35 16.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16.36 έχει καταπέσει ναι. 16.40 16.40 αποχές απορρίπτεται 16.41 ναι παρακαλώ You want me to go back to something? No. Λέτε να επανέλθω σε κάποια? I'm not following. Okay, okay. So, so where we are now? In πού είμαστε. 16.41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 της Επιτροπής Μεταφορών υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1644 υπέρ κατά αποχειριστικτή 1646 υπέρ κατά αποχειριστικτή Κατά πίπτη μάλιστα 108 8 της Ήτρε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1649 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 της Επιτροπής Περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1652 από ψηφίζουμε τη 1652 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1654 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται 1660 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι καλό λέω 1656 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1657 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1661 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1662 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1663 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 148 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 αποσχόληση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1670 ε, υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 1671 υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 1672 υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 1673 υπέρ κατά αποχή απορρίπτεται 552 υπέρ κατά αποχή δεκτή 1676 ε, προφορική τροπολογία είναι κάποιο κατά όχι ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16,79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές δεκτή 150 υπέρ κατά αποχές δεκτή Κοντ 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή Και πάλι εδώ πέρα έχουμε ρύθμιση των χρηματοοικονομικών, δεν την κάνουμε. 1693 στην 306 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1698 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Και μετά 1700 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τώρα πρέπει να επαληθεύσουμε 1721 ε, ψήφισμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1722 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1726 υπέρ κατά 1726 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17-28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Πηδάμε τώρα κάποιες γιατί αφορούν τη ρύθμιση των χρηματοοικονομικών και περνάμε σελίδα τρία, 1-4. 1747 Μανέσκου 1747 υπέρ κατά αποχές δεκτή control 58 υπέρ κατά αποχές δεκτεί 1751 υπέρ κατά αποχές απορριπτεται 1752 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1755 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 της απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά συγγνώμη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1766 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1768 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 της ελέγχου Προβλογισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται της Επιτροπής Ελεύθερου απασχόληση 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 1782 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 της απασχόληση υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1787 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 της ανεξοβουλισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1790 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήτρε 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κόντ 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1798 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 1795 1795 υπέρ κατά αποχές απορριφθείτε 1796 υπέρ κατά αποχές απορριφθείτε 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 159 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1802 υπέρ κατά αποχές δεκτή 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή 161 υπέρ κατά αποχές δεκτή 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή 165 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές απορριφθείτε 63 των γυναικών 64. Ε, κόντ 64 υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Και τώρα. Α, 63 τη επιτροπή Γυναικών. Υπέρ κατά αποχέ, απορρίπτεται. Και τώρα έχουμε μία ψήφο για το... Το ΣΥΣΕΦ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το κοινωνικό ταμείο 1807 υπέρ συνεχίζουμε Έχουμε ακόμα δύο λεπτά νομίζω. Συνεχίζουμε. Να συνεχίσουμε, να συνεχίζουμε. 1807 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται.

Κοιτάξτε, συναδελφοί, περνάμε στην 18.08, ε, σελίδα 324. Κοιτάω εγώ. Ε, κοιτάξτε εσείς που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση αγαπητοί συνάδελφοι γιατί πρέπει να ελέγχουμε πολλά πράγματα ε, και το πώς ψηφίσαμε μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω πως είναι καλύτερα να διακόψουμε, να προετοιμάσουμε ε, ε, να τα δει η γραμματεία και τρεις η ώρα ακριβώς παραλαμβάνεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.